Yes, <clears throat> you're absolutely right. It's the one who are in time that should be rewarded. Βεβαίως, ε, καλημέρα σας. Δεν πρέπει να τιμωρήσουμε αυτούς που ήρθαν στην ώρα τους. Καλημέρα σας ε, για την ε, δεύτερη μισή μέρα συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Εγκρίνουμε τη μέση διάταξη αν δεν έχετε προτάσεις τροποποίησης. Έχουμε δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο είναι η παρουσίαση της έκθεσης από τους δύο μας και μετά θα ακούσουμε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από δύο χωριστές υπηρεσίες. Όπως ξέρετε, η ενδιάμεση εκθεσή μας ε, με βάση την εντολή της 17ης Δεκεμβρίου η Επιτροπή μας πρέπει να υποβάλει ενδιάμεση έκθεση. Όπως όλοι γνωρίζετε, οι συντονιστές συμφώνησαν να γίνει σε αποκλειστικά τεχνική βάση να δώσω το λόγο στον κύριο Φάλβα. Ευχαριστώ αγαπητή Πρόεδρε. Εδώ και πάνω από έξι μήνες το Κοινοβούλιο αποφάσισε να συσταθεί αυτή η Επιτροπή Έρευνας για να ερευνήσουμε τις ε, κατηγορίες ότι δεν εφαρμόστηκε σωστά το ενωσιακό δίκαιο σε σχέση με τη μέτρηση των καυσαερίων των αυτοκινήτων. Όπως όλοι γνωρίζετε, αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση την εντολή μας, οι έρευνες, οι έρευνες μας πρέπει να στοχεύουν στην ε, υποχρέωση τήρησης των κανόνων, στον ε, κανονισμό για τα όρια των ε, εκπομπών των αυτοκινήτων. Είναι ένας κανονισμός του 2007. Επιπλέον, πρέπει να συλλέξουμε πληροφορίες για να δούμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη έχουν στοιχεία για τη χρήση αυτών των μηχανισμών αλλίωσης και επίσης συλλογή στοιχείων για το κατά πόσον έχει ε, εφαρμοστεί η οδηγία 46 του 2007. Συναντηθήκαμε με πρόσωπους του κλάδου, μηχανικούς, ε, περιβαλλοντολόγους και κάποιους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής και τον Σεπτέμβριο και όπως ξέρετε το Σεπτέμβριο ακούσαμε τους επιτρόπους και ε, για να μας πούν τι έκαναν και, και λυπάμαι που ο κύριος Φερχόγεν είναι κρίμα που δεν θέλησε να παρευρεθεί αλλά παρόλα αυτά πρέπει να ευχαριστήσουμε την πρόεδρό μας που επέμεινε από αυτήν την άποψη, συγγνώμη, τον προσεχή Σεπτέμβριο. Λοιπόν, Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Σε αυτήν την ενδιάμεση έκθεση που σας υποβάλλουμε σήμερα αποφασίσαμε μέχρι στιγμής να μην συμπεριλάβουμε πολιτικά συμπεράσματα γιατί είναι ενδιάμεση έκθεση. Θεωρούμε ότι σε αυτή τη φάση είναι πρόωρο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλύτερη αξιολόγηση για το τι συνέβη και μια καλύτερη εκτίμηση γιατί ακριβώς είναι Ποια είναι η αλήθεια. Είμαι στην ε, διάθεσή σας για να ακούσω τα σχόλιά σας. Και τώρα ο συνάδελφος ε, συνεισηγητής, τον οποίο δεν βλέπω, είμαι σίγουρος ότι θα θέλει να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κερμπράντη, θέλετε να μιλήσετε τώρα ή στο τέλος. Α, στο τέλος, ωραία. Οπότε να, μιλήσουμε, να μιλήσουν τώρα Ευχαριστώ. Ε, οι σοσιαλδημοκράτες, λέει εκπρόσωπος των σοσιαλδημοκρατών, ε, στηρίζει αυτήν την ε, έκθεση που απλώς αποτυπώνει την κατάσταση πρόοδου γιατί κάναμε ήδη κάποιες πρώτες ακροάσεις που καταδεικνύουν πόσο σκόπιμη ήταν η σύσταση αυτής της Επιτροπής Έρευνας. Σε αυτό το στάδιο δεν έχω περισσότερα διότι είναι απλώς ενδιάμεση έκθεση και φυσικά θέλω να συνεργαστούμε με τους δύο συζητητές για την τελική έκθεση και είμαι στη διάθεσή τους. Ευχαριστώ. αυτό του μηχανισμού αλλίωσης το συγχαίουμε με τις διαφορές εκπομπών μεταξύ κέντρου ελέγχου και πραγματικών συνθήκων οδήγηση. Δεύτερον, ορισμένοι εμπειρογνωμόνες προσκλήθηκαν για να παρουσιάσουν τις ιδεολειπτικές τους απόψεις που δεν έχει να κάνει με την εργασία της Επιτροπής μας. Και τρίτον, δεν νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία ότι η τεχνολογία των κινητήρων diesel δεν μπορεί να τηρήσει αυτά που θα θέλαμε να τηρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Χένκελ, ο κύριος Ηλικιώτης. Α, δεν είναι παρόν. Ο κύριος Έκχοντ. Είναι έξω. Είναι έξω. Ίσως θα έρθει, λέει ο ο κύριος Ηλικιώτης από τη δική μας οπτική γωνία. Ευχαριστούμε τους συζητητές Μόνο μία παρατήρηση. Μέχρι τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επικριτικοί για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμεθα με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, τι έγραφα μας δίνουν, πώς απαντούν τις ερωτήσεις μας, τι πρόσβαση μας δίνουν σε όλη την απαραίτητη πληροφόρηση. Είναι πολύ βραδία αυτή η διαδικασία δεν βλέπουμε να υπάρχει εντό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαρκής καλή βούληση. Και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία μια επιτροπή ακριβώς ε, έρευνα. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολύ επικριτικές και κατηγορηματικές δηλώσεις. Ούτω ή άλλω ε, τα πορίσματα θα είναι στο τέλος, κάτι το οποίο είναι καλό, γιατί υπάρχει πρόοδο. Ελπίζω στο δεύτερο ε, ήμιση της εργασίας μας να υπάρξει ταχύτερη πρόοδο και ιδίω οι υπηρεσίε τη Κομισιόν να καταλάβουν ότι το να μα κρύβουν πράγματα σε τελευταία ανάλυση θα ε, είναι προζημία, ε, προζημία Ευχαριστώ κύριε Συγκητώτη. Ε, πρέπει να πω ότι ε, για αυτόν το ε, η ομάδα μας υποστήριξε από την αρχή ότι έπρεπε να αξιοποιήσουμε αυτή την αρχική έκθεση για να δώσουμε μια πρώτη πολιτική εκτίμηση της υπόθεσης. Ε, άλλωστε έχουμε αρκετά στοιχεία από τις ακροάσεις και από τα γραπτά κείμενα που μας έχουν σταλεί. Ε, κατά άποψή μας αποδεικνύονται και ευθύνες της Κομισιόν αλλά και των κρατών μελών για αυτό το σκάνδαλο. Ε, εν τούτης, εμείς ε, πιστεύω, αν η πλειοψηφία των ομάδων υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι τεχνικό, πρέπει να παραμείνει στα διαδικαστικά θέματα. Ε, γιατί θεωρούμε ότι η παράγραφος G, όπως διατυπώνεται, ε, εκφράζει και μια πολιτική εκτίμηση. Το ότι μέχρι σήμερα δεν βρήκαμε κάποια στοιχεία. Εμείς θεωρούμε, εάν θα παραμείνουμε σε τεχνικό επίπεδο, τότε πρέπει να αναδιατυπωθεί η παράγραφο G και να είναι ακριβώς να εκφράζει μόνο των τεχνικών επίπεδων. Ότι μέχρι τώρα κάνουμε μια ε, ε, ε, αρχική έκθεση και παραμένουμε μόνο στα διαδικαστικά. Και ε, είναι γι' αυτό που εμείς στηρίζουμε την, να υπάρξει διόρθωση σε αυτήν την παράγραφο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Um, the floor to Mr. Gerbrandi, who will address the issues also on paragraph G, I think. Mr. Gerbrandi. Yes, um, thank you very Madam and let, me start ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή τον κύριο Θάλμπα και την γραμματεία της Επιτροπής, της Επιτροπής και τους συναδέλφους για τη συνεργασία που μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε αυτή την ενδιάμεση έκθεση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι μια έκθεση, η οποία απλώ αναφέρεται διαδικαστικά. Όσον αφορά τώρα την παράγραφο G, εγώ πιστεύω ότι και αυτή, όπω έχει διατυπωθεί, αναφέρεται στα διαδικαστικά. Εμείς ω Εξεταστική Επιτροπή θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα στο τέλος ε, των εργασιών μα. Θα ήταν πρόωρο να ε, διατυπώσουμε από τώρα ενδιάμεσα συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, ε, θα ήθελα επίσης να ασκήσω και κάποια κριτική. Κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ήδη από τις 7 Απριλίου και από τις 14 Απριλίου οι συντονιστές είχαν εγκρίνει τη, να, υποβληθούν αιτήματα εγγράφων, υποβολής εγγράφων από την ε, επιτροπή και ακόμα δεν τα έχουμε λάβει. Έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από, τις, από τα μέσα Απριλίου. Αυτό είναι υπερβολικά μεγάλος, μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδίω αν λάβουμε υπόψη μα ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα έχει διάρκεια ζωή 12 μήνε. Το να χρειάζεται να περιμένουμε δύο μήνε για να λάβουμε τα έγγραφα είναι υπερβολικό. Να σα δώσω ε, ένα παράδειγμα. Στη χώρα μου, στην Ολλανδία, στη χώρα μου, δεν ξεκινάει τις εργασίες της μια εξεταστική επιτροπή αν δεν έχει ακόμα λάβει όλα τα έγγραφα που ζήτησε. Εμείς αναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε τις ακροάσεις πριν ακόμα να έχουμε λάβει τα έγγραφα που απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτός βέβαια των ε, ήδη δημοσίων, δημοσίων προσβάσιμων γράφων. Το θεωρώ αυτό παράδεκτο. Πραγματικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και βεβαίως όταν ζητάμε έγγραφα δεν περιμένω να τα λαμβάνουμε σε 24 ώρες. αλλά εγκαίρος. Και θα ζητήσω λοιπόν, θα πετήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να είναι πιο συνεργάσιμη την προηγούμενη εβδομάδα στις ε, κάτω χώρες στην Χάγη το Κοινοβούλιο οργάνωσε μια συνέντευξη τύπου όπως γίνεται τακτικά κάθε λίγες εβδομάδες ε, μέλη του Κοινοβουλίου καθώς επίσης και ε, μέλη της κυβερνήσεως δίνουν τις, ε, μια, μια, μια ουδέτερη ε, ενημέρωση στους δημοσιογράφους και με εκπρόσωπο μάλλον και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτή τη φορά λοιπόν, αυτή την τελευταία εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να παρευρεθεί. Αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Δεν ξέρω εάν κρύβεται κάτι πολιτικό από πίσω, αλλά μου βρωμάει. Και θα ήθελα να ζητήσω για άλλη μια φορά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, συνεργαστεί ως οφείλει, να αποστείλει τα έγγραφα που έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα οποία ε, θα συμβουλευτούμε ε, τηρώντας πλήρως τους κανονισμούς ασφαλείας επίσης. Αυτά είχα να πω, ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους ε, για τη συνεργασία που έχει οδηγήσει σε ομαλή και παραγωγική διεξαγωγή των εργασιών της Εξεταστικής μας Επιτροπής. Ε, μπορούμε να εγκρίνουμε την ε, διάμεση έκθεση πιστεύω και να προ, προσδοκώ στη συνέχιση των εργασιών μας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ τους δύο τους ε, συνεισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές για όλη την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο μας κάνει ισόδεξους και για το μέλλον. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα των εγγράφων, θα ήθελα να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης των συντονιστών δίνουμε το μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει ε, όλο και περισσότερο α, ε, εκφράζει την απογοήτευσή της η Επιτροπή μας εξεταστική για το γεγονό ότι δεν έχει λάβει αυτά τα έγγραφα και συνεχίζει να τα απαιτεί η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, οι οποίες φαντάζομαι δεν θα είναι πολλές είναι αύριο ε, μεθαύριο μάλλον, 22 Ιουνίου, στις 6 το απόγευμα. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 13 Ιουλίου του 2016 και για την... θα συζητηθεί η ενδιάμεση έκθεση στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις μπορούμε να συνεχίσουμε με την ακρόαση. Είναι κάπως ιδιαίτερη η ακρόασή μα σήμερα. Έχουμε τέσσερις εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκ των οποίων ο ένας, όχι δύο, ο ένας, έχει συνταξιοδοτηθεί. Θα του παρουσιάσω. Ο... Στα αριστερά μου κάθεται ο κύριος Βένολε Κοζίκο. Από τον Ιούνιο του 2015 ήταν υπεύθυνο για την οικονομική ανάλυση στην ε, αρμόδια γενική διεύθυνση της Επιτροπής. Μετά η κυρία Ιωάννα Σικόφσκα, ε, είναι η σημερινή διευθύντρια της μονάδας για την αυτοκινητοβιομηχανία από το 2015 μέχρι σήμερα. Ε, ο κύριος Φιλιπ Ζαν, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος διευθυντής της σχετικής μονάδας από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι το 2015 και ο κύριος Ράινχαρτ Σούλτε Μπράουξ Διευθυντή τη ίδια μονάδα, αλλά μέχρι το Δεκέμβριο του 2007. Έχουν σημασία αυτές οι χρονικές περίοδοι που σας ε, είπα για να ξέρουν τα μέλη της Επιτροπής αν θέλουν να ρωτήσουν κάποιον από τους ε, εκπροσώπους ε, της Επιτροπής μια συγκεκριμένη ερώτηση για ποια χρονική περίοδο ήταν υπεύθυνο ο, καθένα. καθένας. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κοζιγκού ο οποίος είναι στην Γενική Διεύθυνση Grow, θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί η διαδικασία της επιτροπολογίας, ε, την σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας της TCMV, Τεχνικής Επιτροπής για τα ε, Αυτοκίνητα. Και επίσης θα μας εξηγήσει πώς αυτή η Επιτροπή εξέτασε τις, ε, τους ελέγχους δοκιμή, ε, τους ελέγχους σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, τα, το RD. Επίσης θα μας ε, εξηγήσει τη σύνθεση και την λειτουργία της TAAEG, ε, της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τις Συγκρίσεις Τύπου. Έχουμε χρόνο πολύ στη διάθεσή μας, αρκετές ώρες για να ε, τεθούν ερωτήματα. Ω ήθιστε θα δίνουμε από το λόγο πρώτα στους ε, εισηγητέ, μετά στου εκπροσώπους των πολιτικών των ομάδων και του Σκιώδη. Θα ήθελα να ζητήσω από του συναδέλφου, όταν θέτουν ένα ερώτημα να λένε προ ποιον από του τέσσερι εκπροσώπου τη Επιτροπής απευθύνεται. Κύριε Κουζίγκου, έχετε το λόγο για 20 λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί αντιπρόεδροι, αγαπητά μέλη, κυρίε και κύριοι, Χαίρομαι που μας προσκαλέσατε και τους τέσσερις σε αυτήν την ε, ακρόαση σήμερα όπως μου ζητήθηκε. <clears throat> Θα μιλήσω στην ε, εισαγωγή μου για τα δύο αυτά συμβουλευτικά σώματα που οι δραστηριότητε του έχουν να κάνουν με την εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων οχημάτων. Λειτουργούν σε διαφορετικό πλαίσιο και με διαφορετικού στόχου. <clears throat> Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διευκρινίσω τα καθήκοντα, τη σύνθεση και τον τρόπο εργασίας της Τεχνικής Επιτροπής για τα οχήματα, αυτοκίνητα οχήματα, TCMV, και στη συνέχεια θα εξηγήσω πώς η διαδικασία της αγωγής των ε, δοκιμασιών σε πραγματικές συνθήκες του RDA αντιμετωπιστήκε από την TCMV και επίσης θα αναφερθώ στο ρόλο της Κομισιόν και, και των κρατών μελών στην ομάδα ε, εμπειρογνωμόνων για, τον, για την έγκριση τύπου TAAEG και θα δείξω ποιε είναι και οι διαφορέ μεταξύ αυτή τη ομάδα εμπειρογνωμόνων και τη TCMV. Ξεκινώ με την TCMV, την Τεχνική Επιτροπή για τα Αυτοκίνητα Οχήματα. Η TCMV λειτουργεί με του κανόνε τη λεγόμενη επιτροπολογία. Οι συνδίκες προβλέπουν ότι η πρωτογενή ευθύνη για την εφαρμογή τη νομοθεσία είναι στα χέρια των κρατών μελών. Όταν όμω είναι απαραίτητο να υπάρχουν ενιαίε συνθήκε εφαρμογή για την νομοθεσία, μια νομική πράξη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εκχωρήσει εκτελεστικέ εξουσίε στην Κομισιόν. Η Κομισιόν για να μπορέσει να φέρει σε πέρα αυτό το εγχείρημα που την επιφορτίζουν οι συνομοθέτε, πρέπει να αναπτύξει τα εφαρμοστικά μέτρα σε συνεργασία με μια επιτροπή όπου συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη. Γενικά, οι εμπειρογνώμονε, οι οποίοι εκπρόσωπουν τα κράτη-μέλη τη Επιτροπή, έχουν διοριστεί από τις ε, αρχές τους, τις εθνικές αρχές και έχουν την ε, εντολή να εφαρμόσουν την άποψη της χώρας τους σε κάθε σημείο το οποίο τίθεται σε συζήτηση. Η εσωτερική συζήτηση και ο καθορισμός θέσεων μεταξύ των διαφόρων φορέων γίνεται σε εθνικό επίπεδο. Επομένω, πρόκειται για μια διαδικασία μέσα από την οποία τα κράτη-μέλη ελέγχουν την ε, παράγωγη νομοθεσία, της, μάλλον της, ε, αρμοδιότητες παράγωγης νομοθεσία της Κομισιόν όταν διατυπώνει εφαρμοστικές πράξεις. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες οι οποίες είναι δυνατέ, Η επιλογή γίνεται από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σε κάθε πράξη συναπόφασης και λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστεί το είδος της πράξης, το είδος των εφαρμοστικών εξουσιών που εμπλέκονται. Επί τη βάση της διαδικασίας λοιπόν που αναφέρεται στην πράξη της συναπόφασης, οι γνωμοδοτήσεις του είναι ε, οι θέσει των συνομοθετών είναι δεσμευτικέ για την Κομισιόν. Η νομοθεσία για, τα, για τι εκπομπέ των οχημάτων έγινε το 2007 και επομένω η διαδικασία αυτή που εφαρμόζεται είναι η ρυθμιστική, η κανονιστική διαδικασία με δυνατότητα ελέγχου. Η συνθήκη τη Λισαβόνα έχει εισαγάγει τροποποίηση στην Επιτροπολογία, αυτό ελαμβάνει και τη διάκριση μεταξύ εφαρμοστικών και κατεχώρηση πράξεων που ετέθησε ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2009. Αυτές οι πράξεις δεν εφαρμόζονται ακόμα Πλήρω στην ε, νομοθεσία περί έγκριση τύπου. Μια διαδικασία συναπόφαση η οποία θέλει να εναρμονίσει με τη συνδίκη τη Λισαβόνα αυτή τη νομοθεσία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον των συνομοθετών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η TCMV είναι λοιπόν μια κανονιστικού χαρακτήρα επιτροπή μέσα στο πλαίσιο της επιτροπολογίας. Ώστε αυτή εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και έχει εκπροσώπηση των κρατών μελών και προεδρεύεται από την Κομισιόν. Η TCMV δίνει γνωμοδοτήσεις για τα εφαρμοστικά μέτρα τα οποία προτείνονται από την Κομισιόν επί τη βάση μιας ειδικής πλειοψηφίας. Για την κανονιστική διαδικασία μεταελέγχου, η οποία είναι η εφαρμοζόμενη επιτροπολογική διαδικασία, είναι απαραίτητη η θετική γνώμη της Κομισιόν για να μπορέσουν να εγκριθούν τα προτινόμενα εφαρμοστικά μέτρα. Τα εφαρμοστικά αυτά μέτρα θα πρέπει να περάσουν τον έλεγχο και του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Τούτων λεχθέντων. Ας εστιάσω στο πακέτο μέτρων για τις πραγματικές εκπομπές ε, των οχημάτων στον δρόμο και τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίσαμε. Θέλουμε να έχουμε διαδικασίες οι οποίες να είναι ε, στεναρές και ατεκτικές για την για τον έλεγχο των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκε οδήγηση. Αυτό βασίστηκε στις μελέτες που έγιναν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η αρχική τεχνική εργασία έγινε από την Ομάδα Εργασίας για τις Πραγματικές εκπομπέ σε φάση οδήγησης των ελαφρών οχημάτων η οποία ε, ομάδα έδωσε τεχνογνωσία και τεχνική αρρωγή στην Κομισιόν. Ο στόχο είναι να υπάρχει αυτή η νέα διαδικασία RDE, η οποία να λειτουργεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2017, όπω ανακοινώθηκε από την Κομισιόν το 2012 στην ανακοίνωσή τη CARS 2020. 1η Απριλίου 2014 η Κομισιόν παρουσίασε στα κράτη-μέλη μέσω τη TCMD την, ε, το όραμά τη για την αρχιτεκτονική αυτού του πακέτου RDE. Αυτό ε, ε, επικυρώθηκε και από την νομοθεσία για τα Euro 5 και 6 οχήματα, η οποία είναι ο κανονισμός 715-2017. Η Κομισιόν παρουσίασε ένα οδικό χάρτη, ο οποίος προτείνει η νομοθεσία για τις πραγματικές ε, εκπομπές να βρίσκεται σε τέσσερα νομοθετήματα, τα οποία δεν θα προχωρήσουν όλα με την ίδια ταχύτητα. Η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν είναι εφικτή από τεχνική και διοικητική άποψη και έγινε δεκτή από τα κρατημέρια στην TCMV. Αλλά επειδή κάθε ένα από τα νομοθετικά κείμενα θα έπρεπε να εγκριθεί από μια ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος καθυστερήσεων. Οι συζητήσει για το αντί εισήχθησαν στην ατζέντα των επομένων συναντήσεων της TCMV στο διάστημα Απριλίου 2014 με Μάιο 2015. Δέκα περίπου συναντήσεις. Δεδομένου επίσης του γεγονότος ότι η ανάπτυξη της διαδικασίας δοκιμασιών κάτω από πραγματικές συνθήκες σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των οξυδίων του αζότου, περιελήφθη αυτό το τμήμα στο πρώτο σχέδιο για την πρώτη, στο σχέδιο για την πρώτη πράξη σε σχέση με το ΑΝΤΙ. Ο κανονισμό αυτό ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο, διότι έπρεπε να λάβει υπόψη από τη μια πλευρά τον νομικά ορθό τρόπο εφαρμογή των κανόνων για τα όρια εκπομπών σε κάτω από φυσιολογικέ συνθήκες όπω αναφέρεται από τον κανονισμό Euro 5-6 και επίσης τα, τις ανησυχίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων οξυδίου του αζότου. Επίσης όμως θα έπρεπε να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των αυτοκινητοβιομηχανιών. Μέχρι το τέλος του 2014 η TCMV είχε υποστηρίξει γενικά τη διαδικασία δοκιμασίας RDE δηλαδή την ουσία του σχεδίου για τον πρώτο κανονισμό RDE. Αλλά υπάρχουν μερικά στοιχεία τα οποία είναι ακόμα υπό συζήτηση μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να τροποποιηθούν. Οι συζητήσει που έλαβαν χώρα μετά το Νοέμβριο του 2014 εστίασαν περισσότερο στι ε, ενδείξει σε αιτιολογικέ σκέψει των περαιτέρω προθέσεων τη Κομισιόν για το δεύτερο νομοθέτημα, RDE. Τα κύρια θέματα είναι ο ορισμό των συμπληρωματικών οριακών συνθήκων και τα ρυθμιστικά όρια τα οποία δεν πρέπει να, ε, το οποίο δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση, τα λεγόμενα NTE, not to exceed, τα οποία εφαρμόζονται σε αυτές τις δοκιμασίες. Τα όρια αυτά, τα NTE, επιτυγχάνονται με το να πολλαπλασιάσει κανεί το όριο που βρίσκεται στον κανονισμό με τους παράγοντες της συμμόρφωσης. Αυτά δεν έχουν καμιά σχέση με την πρώτη πράξη αντί. Μετά από την διαβούλευση μεταξύ όλων των υπηρεσιών της Κομισιόν, το σχέδιο κανονισμού περιελήφθη στην ε, ημέρησια διάταξη της TCMV στις 24 Μαρτίου 2015 για να μπορέσει να γνωμοδοτήσει η TCMV. Δυστυχώ όμω, σε αυτή τη συνάντηση, μετά από ένα πρώτο γύρο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών, δεν υπήρξε δυνατότητα εξέβρεση μιας ειδική πλειοψηφία. Και πριν από τη συνάντηση πράγματι αυτή, η Γερμανία είχε υποβάλει μια πρόταση συμβιβασμού η οποία δεν περιλάμβανε ημερομηνίε στόχου για την εισαγωγή των παραγόντων συμμόρφωση και πρότεινε να εφαρμοστούν αυτοί οι παράγοντε σε δύο φάσει μέσω μια αιτιολογική σκέψη. Λόγω τη ε, ε, υποβολή αυτή τη πρόταση την τελευταία στιγμή, αυτό δεν μπορούσε να γίνει δεκτό από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη γιατί δεν είχαν συμμετεί στη θέση του σε σχέση με αυτή την πρόταση. Γι' αυτό η γνωμοδότηση τη CMV για το σχέδιο τη πρώτη ε, πράξης RDE ψηφίστηκε στην επόμενη συνάντηση 19 Μαΐου 2015 από μια πλειοψηφία των παρόντων κρατών μελών. Αμέσως μετά την πρώτη ρυθμιστική αυτή πράξη και την έγκρισή της, η Κομισιόν υπέβαλε το σχέδιο για την δεύτερη ρυθμιστική, κανονιστική μάλλον πράξη RDE, η οποία ανακρίθηκε από τη CMV 28 Οκτωβρίου 2015. Η, το σχέδιο αυτό κανονισμού προκύπτει από την ε, ανάλυση των αβεβαιοτήτων που έχουν να κάνουν με τα κινητά συστήματα μέτρησης ε, εκπομπών, τα PEMS, και επίσης επί τη βάση των δεδομένων που έχουν αποκτηθεί από τα τωρινά συστήματα PEMS. Η δεύτερη νομοθετική πράξη λοιπόν αφορά τους ποσοτικούς στόχους για τα οξύδια του αζότου κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών RDE. Αυτό γίνεται με τον καθορισμό των παραγόντων συμμόρφωσης. Αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης καθορίζουν τα μέγιστα επίπεδα εκπομπών σε όλες τις δυνατές συνθήκες του κύκλου δοκιμασιών και αυτό περιλαμβάνει και τις ανοφέρειες. Άρα είναι υψηλότερα αυτά τα όρια από τους όρους του κανονισμού 5-6 που καθορίζει τις μέσες εκπομπές. Ο, η δεύτερη κανονιστική πράξη RDE εισάγει επίσης την υποχρέωση για τους κατασκευαστές να δηλώνουν τη στρατηγική του για των εκπομπών. Το αρχικό σχέδιο της Επιτροπής ήταν πολύ φιλόδοξο γιατί ε, πρότεινε παράγοντες ε, συμμόρφωσης στην χαμηλότερη, ε, στο χαμηλότερο όριο της κλίμακας του φάσματος με βάση την νομική και τεχνική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά χρειάστηκε να τροποποιηθεί για να εγκριθούν, για να πάει προς υψηλότερους παράγοντες συμμόρφωσης αν και πάντα μέσα στο φάσμα ούτως ώστε να υπάρξει ειδική πλειοψηφία μεταξύ των κρατών μελών και οι παράγοντες συμμόρφωσης που ψηφίστηκαν συνολικά, τελικά, είναι στα πλαίσια του φάσματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασιζόταν στην τεχνική ανάλυση. Σε αυτή τη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για την τρίτη και την τέταρτη ρυθμιστική πράξη RD. E η τρίτη θα υποβληθεί ακόμη φέτος, ενώ η τέταρτη αναμένεται στις αρχές του 2017. Η τρίτη θα καθορίσει τη διαδικασία για τη μέτρηση των σωματιδίων και θα συμπεριλάβει και το αποτέλεσμα της ε, αρχής λειτουργίας των κινητήρων σε κρύες συνθήκες. Και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δημοσιεύουν τους παράγοντες συμμόρφωσης για κάθε αυτοκίνητο στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Έτσι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τις πραγματικές εκπομπές. Τέλος, στην τέταρτη ρυθμιστική πράξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καθορίσει τους κανόνες για ανεξάρτητη μέτρηση RD όταν τα αυτοκίνητα είναι εγκινήσει συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμιστικών επιπτώσεων εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση. Για να καταλήξω για τη διαδικασία RDE, να αναφέρω ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, η πρώτη διαδικασία τεστ RDE έγινε με βάση τις μελέτες που έγιναν από το Κοινό Κέντρο Έρευνων ε, και την προπαρασκευαστική εργασία τεχνικών εμπειρογνωμόνων σε στην ομάδα εργασία για τι πραγματικέ εκπομπέ ελαφρών οχημάτων. Αυτή, η ομάδα εργασία λέγεται RDELDV. Δεύτερον, τα θέματα που τέθηκαν στη συζητήσει του TCMV εκτιμώνται προσεκτικά από τι υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά και επιστημονικά στοιχεία και μεταφέρονται για τεχνική συζήτηση στην ομάδα εργασία RDELDV αν χρειάζεται. Τρίτον, η διαμόρφωση συνένεση και η δυνατότητα να επιτευχθούν συμβιβασμοί είναι ζωτική για να εγκριθούν εγκαίρως ε, τα, οι προτάσεις ε, εφαρμοστικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι στην Επιτροπή αυτή τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να μπλοκάνουν τη διαδικασία. Επίσης, επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε αυτήν την ε, δυνατότητα δημιουργίας συνένεσης, διότι τα κράτη-μέλη στην σχετική επιτροπή μπορούν να μπλοκάρουν μια πρόταση γιατί χρειάζεται ειδική πλειοψηφία για να περάσει μια πρόταση. Τέταρτον, παρά το ότι υπήρξε μια ελαφρή καθυστέρηση για την έγκριση της πρώτης πράξης RDE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι καθυστέρησε η ψηφοφορία στο TCMV, αυτό δεν επηρέασε το χρονοδιάγραμμα που προβλεπόταν από την αρχή για αυτή τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα απέδε μεγάλη σημασία στην έγκαιρη πρόοδο του θέματος αυτού και θεωρούσε ότι η απόφαση RDE είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας. Η διαδικασία Test RDE ήδη έχει αρχίσει να ισχύει για λόγους επιτήρησης από τις αρχές του 2016 και σε εφαρμοστεί μαζί με τους παράγοντες συμμόρφωσης από το Σεπτέμβριο του 2017. Τέλος, θα πω δύο λόγια για την ομάδα εμπειρογνωμόνων έγκρισης τύπου. ΤΑΕΚ είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου συμμετέχουν διάφορες εθνικές αρχές εγκρίσης τύπου, λειτουργεί ε, με άτυπο τρόπο και δεν παίρνει δεσμευτικές αποφάσεις, αντίθετα από το TCMV. Δημιουργήθηκε το 2010 για να διασφαλίσει διαφάνεια και την αναγκαία ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και των Εθνικών Αρχών Έγκρισης Τύπου. Αυτή η ομάδα TAG προεδρεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι μια πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό ανάμεσα στι εθνικέ αρχέ ε, έγκριση τύπου ούτω ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή τη σχετική νομοθεσία παντού στην Ένωση. Οπότε, ο στόχο του GAAG δεν είναι να παίρνει αποφάσει καθόλου, αλλά αντίθετα προσπαθεί να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών για την ερμηνεία των κανόνων και την εφαρμογή των κανόνων και τα πρακτικά τη είναι στον ιστότοπο τη Κομισιόν και οι ερωτήσει για συζήτηση από το ΤΑΕΚ τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη-μέλη συνήθως μετά από συζήτηση στην Επιτροπή των Αρχών Έγκριση Τύπου, όπου δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με την εργασία της TAG για τις εκπομπές να τονίσω τα εξή δύο. Πρώτον, το χάσμα μεταξύ των τεστ εργαστηρίου και των τεστ πραγματικών συνθήκων για τα οχήματα δεν έχει ζητηθεί στο TAG, γιατί αυτό το αντιμετωπίζει το TCMV. Η εισαγωγή ενός πιο αντιπροσπευτικού κύκλου τεστ, WLTP, και ε, πραγματικών εκπομπών είναι εφαρμοστικά μέτρα που πρέπει να εγκριθούν μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας. Δεύτερον, η χρήση των μηχανισμών αυτών αλλίωσης δεν συζητήθηκε στο TAG πριν από τις αποκαλύψεις για το Volkswagen, για την Volkswagen. Δεν είχαμε καμία αρχή έγκρισης τύπου που να έχει ζητήσει διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ενωσιακά μέτρα για αυτά τα θέματα ή καμία αποστολή στοιχείων για τη χρήση μηχανισμών αλλίωσης που απαγορεύονται από τον ενωσιακό νόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοζίγκο. Θα περάσουμε τώρα στη διαδικασία των ερωτήσεων, ξεκινώντας με τους συζητητές μας. Κύριε Σάρπα. Σάλπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Κοζίλια για τις εξηγήσεις που δώσατε. Χθες ένα βρετανικό έντυπο επέμεινε ότι το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γνώση του γεγονότος ότι κάποιες βιομηχανίες χρησιμοποιούσαν τις συσκευές αποφυγής μέτρησης των εκπομπών. Ένα μέλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών που ήταν εδώ της Επιτροπής είπε σαφώς ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο δοκιμάστηκε έδειξε πάρα πολύ υψηλές ε, εκπομπές διοξιδίου, οξυδίων του αζότου σε χαμηλές θερμοκρασίες και ανήκε στην κατηγορία Euro 6. Επειδή αυτές οι εκπομπές δεν ε, ελέγχονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό πρέπει να οφείλεται σε μια στρατηγική που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής για τις χαμηλές θερμοκρασίες θερμοκρασίες. Βάσει του άρθρου λοιπόν αυτό που δημοσιεύτηκε στο Βρετανικό έντυπο το Νοέμβριο του 2014 ο Γενικός Διευθυντής της Envy, DG Envy, κ. Φάλκεμπερκ, έστειλε μια επιτροπή στον κύριο Καλέχα Κρέσπο της ε, Γενικής Διεύθυνσης του Επιχειρήν λέγοντας ότι θα έπρεπε η Γενική του Διεύθυνση να εξετάσει τις τεχνικές αυτές που εφαρμόζουν ορισμένοι κατασκευαστές για τη μείωση των εκπομπών απενεργοποιώντας σε χαμηλές ε, ε, θερμοκρασίες ε, το σύστημα ελέγχου των εκπομπών επειδή το όχημα χρειάζεται περισσότερη ισχύ. Ήταν υποτίθεται ευθύνη λοιπόν ε, αυτών των Γενικών Διευθύνσεων να ειδοποιήσουν και τα κράτη-μέλη για το πρόβλημα αυτό. Θα ήθελα εγώ να ξέρω εσείς ε, θα μπορούσατε να μου πείτε αν η Κομισιόν ήξερε πράγματι ότι υπήρχαν αυτές οι συσκευές απενεργοποίησης του συστήματος ελέγχου εκπομπών από τις ε, κατασκευαστικές εταιρείες αυτοκινήτων, πότε και αν είχε αυτή τη γνώση η Κομισιόν λοιπόν. Δεν είναι καινούριο πράγμα αυτές οι, αυτοί οι μηχανισμοί Είναι κάτι το οποίο το απαγορεύει η νομοθεσία από 2008. Επομένως, τα κράτη-μέλη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν αυτή την απαγόρευση των μηχανισμών αλλίωσης. Επομένως, η ύπαρξη των μηχανισμών αλλίωσης ήταν γνωστή ως γενικό φαινόμενο ε, στα, και στην Κομισιόν και στα κράτη-μέλη. Βέβαια, ε, τονίζω ότι δεν γνωρίζαμε συγκεκριμένη περίπτωση ε, διάπραξης απάτης. Το πρόβλημα είναι ότι οι μετρήσει δεν αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές καυσερίων σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι διαδικασίες μέτρησης και έτσι ξεκίνησε και αυτό, αυτή η προσπάθεια για να γίνονται οι μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες οδηγίες. Το 2011-2013 δημοσιοποιήθηκαν οι σχετικές μελέτες για το RDE της Επιτροπής και το περιεχόμενο αυτών των μελετών έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τα κράτη-μέλη. Η ομάδα ερευνητική έκανε μετρήσεις των εκπομπών και διαπίστωσε ότι οι εργαστηριακοί έλεγχοι ε, δεν μετρούν ε, το, τα οξύδια του αζότου ε, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ωστόσο, σε αυτές τις μελέτες οι μηχανισμοί αλλίωσης δεν δεν αποτέλεσαν αντικείμενο ε, αυτών των μελετών. Γιατί είχαν άλλο αντικείμενο τις και αυτές οι μελέτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση με τη βάση αυτών των μελετών και είναι όλη αυτή η διαδικασία που σας περιέγραψα για την εισαγωγή ε, μετρήσεων σε πραγματικές ε, συνθήκες. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με την βελτίωση του τρόπου διεξαγωγής των μετρήσεων. Θέλει μήπως η συνάδελφος να συμπληρώσει κάτι. Ναι και ευχαριστώ. Αναφερθήκατε σε ένα άρθρο που έχει δημοσιοποιηθεί στην Guardian όπου καταγγέλλεται η χρήση διατάξεων αναστολής. Θα ήθελα να ευκρινίσω ότι αναφέρεται σε βενζινοκίνητο όχημα και ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Πετρελαιοκίνητο μάλλον. Όχι. Βενζινοκίνητο. Το άρθρο αναφερόταν σε συνθήκε στη μέτρηση των οξυδίων του αζότου όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Ε, δηλαδή όταν ξεκινά ο κινητήρας και ο κινητήρας δεν έχει θερμανθεί ακόμα. Ε, έχουμε διαπιστώσει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριφέρεται ορθά μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήματος. Επομένω, σε αυτές τις περιπτώσεις μια διάταξη αναστολή δεν θα βοηθούσε σε κάτι. Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε έγγραφα τα οποία που ήτυχε στην κατοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα οποία διέρευσαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ξεκινήσαμε μία ακρόαση, ενώ δεν έχουμε λάβει ακόμη τα πρακτικά κάποιων συναντήσεων ε, τα οποία ζητήσαμε. Άρα δεν είναι πολύ καλή κατάσταση. Επίσης, ε, στην ομάδα εργασίας RDLTV μας στείλατε ότι συμμετέχουν ορισμένες οργανώσεις. Αλλά δεν μας στείλατε ποιοι συμμετέχουν. Ποιοι εκπροσωπούν κάθε οργάνωση που μας στείλατε ότι συμμετέχει. Θέλουμε παρακαλώ σήμερα αυτό το κατάλογο με του ποιοι συμμετείχαν. Γιατί θεωρώ ότι αυτό θα μας βοηθούσε πολύ. Δεύτερον, Πόσα άτομα, για παράδειγμα, είναι από τον κλάδο, από τι αυτοκινητοβιομηχανίε, σε αυτές τις ε, τακτικέ συναντήσει, 5, 20, 50. Και ποιο είναι ο σχεσμό δυνάμεων, πώς είναι από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Γιατί είδα ότι μόνο κράτη-μέλη, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ολλανδία, Γερμανία, εκπροσωπούν το. Ε, μπορείτε να μα πείτε τίποτα για αυτό την ε, ισορροπία δυνάμεων. Και σύντομα, παρακαλώ. Ε, σύντομα, ναι. Ναι. Το θέμα δεν είναι ποιος ε, μπορεί να συμμετάσχει, αλλά και τον αριθμό για τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν και στις εργασίες του CMV e που είναι ο σωστός τόπος για να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Κάποια κράτη-μέλη ενδιαφέρονται περισσότερο, άλλα λιγότερο. Τώρα, πόσοι συμμετέχουν. Φυσικά, διάφορες οργανώσεις ε, στέλνουν τους ε, εκπροσώπους τους ανάλογα με το δυναμικό τους αλλά ποτέ δεν ήταν 10-20 από ένα φορέα, ενώ οι άλλοι είχαν πολύ λιγότερους. Ευχαριστώ. Παρακαλώ μπορείτε να μας στείλετε την πληροφόρηση. Όχι μόνο ποιοι φορείς συμμετείχαν, αλλά πόσοι από κάθε φορέα. Δεύτερη ερώτηση. Στην ερώτηση 4 είπατε ότι περιμένατε μέχρι το 2011 για να ξεκινήσει η ομάδα εργασίας RDE-LDV γιατί δεν υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα τύπου Euro 5 στην αγορά. Αλλά για τις διαφορές μεταξύ των τεστ και πραγματικής χρήσης για το Euro 3 και 4 ε, είχαμε ήδη διαφορές λοιπόν σημαντικές. Γιατί χρειάζεται να περιμένετε να έχετε αρκετά αυτοκίνητα τύπου Euro 5 Δύο στοιχεία. Ναι, είχαμε κάποιες πληροφορίες για τις διαφορές, για τις τιμές ε, στο εργαστήριο και τις τιμές πραγματικής οδήγησης για τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούσαν. Τα αυτοκίνητα τύπου Euro 4. Αλλά το κείμενο Euro 5-6 έλεγε εκπεφρασμένα, νομίζω στο άρθρο 14, ότι έπρεπε να ελέγξουμε την απόδοση των οχημάτων Euro 5-6 πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης νέας μεθόδου μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες. Τα πρώτα αυτοκίνητα που εισήλθαν στην αγορά υποχρεώνω, ε, συγγνώμη, υπογραμμίζω ότι η υποχρέωση συμμόρφωση ασχεί το 2011 τα νέα αυτά οχήματα άρχισαν να μπαίνουν στην αγορά τέλη 10 αρχές 11. Έπρεπε λοιπόν να περιμένουμε να υπάρχουν αρκετά τέτοια οχήματα για να τα ελέγξουμε, να τα σε συνθήκε πραγματική οδήγηση, όπω όριζε το κανονιστικό πλαίσιο για τα Euro 5-6. Και αυτό ακριβώ κάναμε. Οι εργασίε ξεκίνησαν τέλο του 2006, λέει ο εισηγητή. μόλι μπορέσαμε να έχουμε τα στοιχεία και ήταν ιδιαίτερα τα στοιχεία του σεμιναρίου που επανειλημμένα αναφέρθηκε στι συζητήσει που είχατε με του συναδέλφους από το Κοινό Κέντρο Έρευνας, Γεμπράντι. Αλλά είχαμε μια κρόαση χτε, όπου υπόθηκε ότι οι εμπειρογνώμονε γνώριζαν ότι ο κύκλο ε, τεστ ήταν απόλυτα ξεπερασμένο πολύ πριν το 2011. Γιατί σα πήρε λοιπόν τόσο χρόνο, γιατί δεν κάνατε τα βήματα αυτά νωρίτερα για να βελτιωθεί αυτό ο κύκλο τεστ. Κομισιόν. Δεν υπάρχει καμία ασάφεια όσον αφορά το ότι όλοι και οι υπηρεσίε των Κομισιών γνώριζαν ότι υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών των τεστ στο εργαστήριο και των τιμών των ε, εκπομπών σε πραγματικέ συνθήκε. Ο κύριος στόχος μας λοιπόν ήταν να καθορίσουμε μια αξιόπιστη και καινοτόμο διαδικασία που θα επέτρεπε να μετρήσουμε με πραγματικό τρόπο τις πραγματικές εκπομπές με σωστό τρόπο δηλαδή. Έχετε δίκιο. Τα στοιχεία ήταν στη διάθεσή μας ήδη το 2008, αλλά αφορούσαν τα οχήματα που συμμορφώνονταν με τους κανόνες Euro 4 και το κείμενο, ο κανονισμός για τις εκπομπές 5-6, Euro 5-6, μας υποχρεώνει να μετρήσουμε τις εκπομπές για τα νέα οχήματα, τα οχήματα που θα έπρεπε λοιπόν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις Euro 5-6, ιδιαίτερα για τις μηχανές diesel. Άρα γνωρίζαμε το θέμα, αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι να περιμένουμε να έχουμε επαρκή στοιχεία για να ξεκινήσουν πραγματικά αξιότιστες μελέτες. Και αυτό κάναμε κατά τη διάρκεια των ετών 11 έως 14, οι οποίες εργασίες μας επέτρεψαν να καταλήξουμε σε μια στρατηγική και λοιπόν στον κανονισμό που λέγεται RDOE, ε, δηλαδή πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Και Μπράντι, ωραία. Νομίζω ότι ε, καρκινοβατούμε, αλλά καταλαβαίνω γιατί η Επιτροπή χρειάστηκε τόσο χρόνο. Λοιπόν. Κύριος Κάρινς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βρίσκω κάπως παράδοξο. Ίσως κάποιος μπορεί να μου εξηγήσει εν συντομία πότε η Κομισιόν συνειδητοποίησε ότι οι μετρήσεις των ε, οξυδίων αζότου στους κινητήρες δίζελ αποτελούσαν ένα πρόβλημα. Μια ημερομηνία μπορείτε να μου πείτε, ένα χρόνο, το έτος που το διαπιστώσατε. Ότι είναι οι εκπομπές ε, πρόβλημα ή οι μετρήσεις των εκπομπών ότι δεν ήταν επακριβείς λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Όταν ενεκρίτη η νομοθεσία για τα Euro 5 και Euro 6 το 2007, ήδη αυτές οι πληροφορίες ήταν γνωστές από τους συνομοθέτες. Γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η ειδική εντολή για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε τις ε, συσκευές μέτρησης. Το 2007 ήταν γνωστό ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μια στιγμή να σας διακόψω. Το 2007 η Κομισιόν ξέρει ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από τους κινητήρες δίζελ αποτελούν πρόβλημα. Ωραία. Σύμφωνοι λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ποια ήταν η αιτία του προβλήματος αυτού κατά την άποψή σας, γιατί υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα, υπάρχει κάποιο αίτιο για το πρόβλημα. Αν κατάλαβα καλά το ερωτήματα, η λόγοι ήταν το είδο τη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στου κινητήρε δίζελ. Ο δεύτερο, η δεύτερη πηγή του προβλήματο ήταν οι δυσκολίε μέτρηση των αντικτύπων των ε, εκπομπών όταν γινόταν η έγκριση τύπου των οχημάτων. Πάλι θα σα διακόψω, εάν μου επιτρέπετε. Γιατί δεν μπορείτε να μας πείτε ότι καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε από πού το πρόβλημα. Ναι, Uh, what I'm looking for is Μια απάντηση η οποία δεν είναι ήδη έτοιμη και προδιαγεγραμμένη. Πέστε μου κάτι το οποίο δεν ξέρω ήδη. Οι κινητήρες δίζελ εκπέμπουν περισσότερα οξύδια του αζότου από ό,τι δεν συνοκινητήρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διακόπτει ο κύριος Κάντς. Έχουμε περισσότερους κινητήρες δίζελ στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχουμε περισσότερους κινητήρες δίζελ στην Ευρώπη από τις ΗΠΑ. Θα το εξηγήσω. Λέω, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Έχουμε κινητήρες σε δίζελ γιατί εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακο από του βενζινοκινητήρες και ο στόχος ήταν να μειωθεί το εκπομπή, εκπομπές διοξίδιου του άνθρακος. Γι' αυτό δεν θέλαμε να μειώσουμε τις εκπομπές αυτές. Ενώ στις Ηνωμένες δεν είχαμε επιβατικά οχήματα ουσιαστικά με κινητήρες ε, diesel. Ωραία. Είπατε σαφώς ότι είχαμε προβλήματα με τις εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου γιατί έχουμε diesel στην Ευρώπη και έχουμε diesel στην Ευρώπη γιατί ο στόχος μας ήταν να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακος, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Λοιπόν, προσπαθώντας να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, η Κομισιόν, όσο είχε κατανοήσει ότι υπάρχει η ανάγκη να ζυγίσουμε τις δύο πλευρές, ότι εάν έχουμε δίζελ θα έχουμε και περισσότερο, δηλαδή εκπομπές οξυδίου του αζώτου. Το είχε συνειδητοποιήσει αυτό η Κομισιόν. Αν δείτε τα στοιχεία, λέω, ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν των Οριακών Τιμών, που έχουν εγκριθεί στι κατηγορίε Euro 5, Euro 6, είδατε ότι κάνουμε μια αποφασιστική προσπάθεια να μειώσουμε τι εκπομπέ οξυδίων του αζότου και έχουμε φτάσει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο το οποίο ισχύει στι ΗΠΑ. Υπήρξε λοιπόν η θέληση από την Κομισιόν να μειωθούν οι εκπομπέ οξυδιών του αζότου. Το επεξεργαστήκαμε το θέμα αυτό και δράσαμε γι' αυτό. Εμείς διαβάσαμε τώρα τα αποτελέσματα του εργαστηρίου που έγινε στις το 2010 για τις εκπομπές οχημάτων, πριν από έξι χρόνια σχεδόν λέει ότι δεν έχουν μειωθεί ούτε έχουν μείνει σταθερές τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχουν μειωθεί ουσιαστικά και με την εισαγωγή των κατηγοριών 5 και 6. Οι εκπομπές λοιπόν διοξιδίου του αζότου σχεδόν φαίνεται να έχουν αυξηθεί. Το 2010 έχετε ένα εσωτερικό έγγραφο που λέει ότι μειώνονται οι εκπομπές από τους βενζινοκινητήρες ενώ από τους κινητήρες δίζελ ουσιαστικά ανεβαίνουν οι εκπομπές. Τι κάνατε για αυτό το πράγμα. Εμεί εγκρίνουμε νομοθεσία που λέει ότι πρέπει να μειωθούν οι εκπομπέ, Αλλά τι κάνατε πραγματικά για να επιτευχθεί ο στόχο της νομοθεσίας. Έχετε δίκιο. Η γνώση του προβλήματος υπήρχε το 2010. Το 2007 ξέραμε ότι υπάρχει η διαφορά μεταξύ των εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες και των εκπομπών στο εργαστήριο. Ο στόχος των ε, προσπαθειών του 2010 ήταν ακριβώς να προσπαθούμε να βρούμε ποιο τρόπο μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις μετρήσεις στο εργαστήριο, οι οποίες δεν είχαν οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών όπως είδαμε το 2010 και το σημείο εκκίνησης ήταν αυτές οι εργασίες που έγιναν το 2010 για να ε, αντικαταστήσουμε τις, μελέτε, τις μετρήσεις σε εργαστήριο που δεν ήταν ικανοποιητικές γιατί δεν οδηγούσαν σε πραγματική μείωση των εκπομπών ανεξάρτητα από αυτά που είχαν γίνει με τις ε, μετρήσεις στο εργαστήριο, να αντικαταστήσουμε αυτή τη μέθοδο εργαστηρίου με μια νέα μέθοδο που θα επέτρεπε να υπάρχει πραγματικός αντίκτυπος στις εκπομπές οξυδιών του, ε, του αζότ. Κύριε Μπονιφά, ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος που ακούσαμε πριν από εσά είπε από το 2004 είχε δια, δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της κάποια στοιχεία για τα, την, τον αντίκτυπο των οξυδίων του αζότου από τους, από τους κινητήρες δίζελ. Το ξέρατε αυτό λοιπόν από το, από το 2004 φαντάζομαι. Επίσης εγώ σοκάρομαι αρκετά όπως και οι συναδελφοί μου και κατανοώ βέβαια ότι υπάρχουν πολιτικά προβλήματα. Κατανοώ ότι υπήρξε μια καθυστέρηση για να υπάρξει μια, προσ... μια συμφωνία των κατών μελών για να προχωρήσουμε στις μετρήσεις πραγματικών εκπομπών RDE. Όπως ξέρετε έχουμε 10.000 πρόωρους θανάτους λόγω των οξυδίων του αζότου. Αυτό δεν είναι κάτι το αμεληταίο. Θα ήθελα λοιπόν να καταλάβω καλύτερα μαζί σας. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν σημεία αντιφατικά στις απαντήσεις σας στα σημεία 4 και 6 σε σχέση με τις συσκευές της διατάξης αναστολής. Λέτε σε ένα σημείο ότι δεν ξέρατε ότι υπήρχατε αυτές οι συσκευές, αλλού λέτε ότι φανταζόστε ότι υπάρχει υποψία χρήσης τέτοιων συσκευών. Μήπως μπορείτε να είστε λοιπόν πιο σαφείς σε σχέση με τη γνώση που είχατε για την ύπαρξη των διατάξεων αναστολής. Ξεκινώ από το τελευταίο για τις διατάξεις αναστολής. Είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό ότι υπήρχε ο ε, κίνδυνος χρήσης ε, τέτοιων διατάξεων, γι' αυτόν τον λόγο απαγορεύονταν και στην νομοθεσία. Απαγορευόταν η χρήση διατάξεων αναστολής. Επομένως αυτό που ήταν γνωστό ήταν ο κίνδυνος. Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν οι συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης διατάξεων αναστολής. Και τέτοιες περιπτώσεις ήρθαν ε, στη, στη, τις μάθαμε τέλος Σεπτεμβρίου με το σκάνδαλο που δημοσιοποιήθηκε. Όμως το ότι υπήρχε ο κίνδυνος ήταν γνωστό και γι' αυτόν τον λόγο προβλεπόταν η απαγόρευση στην ομοθεσία και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όμως την αξιολόγηση ενδεικτύπου του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, αναθεώρηση της οδηγίας 35 ε, του 2003 αναφέρεται ρητά ότι, αυτές, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος χρήσης διατάξεων αναστολής και συστημάτων τα οποία ε, βελτιώνουν την, οδηγική, την, τη συμπεριφορά του, του, του αυτοκινήτου, ότι υπάρχει κίνδυνος χρήσης τέτοιων διατάξεων αυτός ο κίνδυνος αναγνωρίζεται το 2003, όχι το 2015. Το 2013. Συμπληρώνω τον συνάδελφο. Υπήρχε διαρκής ανησυχία για αυτές τις διατάξεις. μια ανησυχία την οποία την είχαμε διαρκώς καθώς συζητείται το σύστημα ε, μετρήσεων σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί είναι δύσκολο να εντοπιστεί μια τέτοια διάταξη. Επομένως, ψάχναμε έναν τρόπο μέτρησης ε, που να μην μπορεί να αλλοιωθεί. Επομένως, αυτή, αυτό που ήταν γνωστό ήταν ο, ο κίνδυνος, η ύπαρξη του κινδύνου ερώτηση. Όμως εδώ δεν συζητάμε για μια αόριστη ανησυχία. Αναφέρεται στην αξιολόγηση αντικτύπου ρητά ότι χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα. Απάντηση της Κομισιόν. Αυτό που διαπιστώναμε επί χρόνια είναι ότι υπήρχε ο κίνδυνος, αναφέρθηκε το 2010, όταν ξεκίνησε η διαδικασία για το RTE, Υπάρχουν αναφορές σε τέτοιες διαδικασίες, σε, σε τέτοιες διατάξεις μάλλον, από το 2010. Υπάρχει σχετική έρευνα του 2013. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε ευαισθητοποιηθεί και γνωρίζαμε τον κίνδυνο χρήσης τέτοιων διατάξεων. Αλλά δεν είχαμε απτές αποδείξεις ότι ε, μία διάταξη αναστολής είχε χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένη περίπτωση. γνωρίζετε την συνάντηση του κυρίου Τάνκερ και και ε, τι γνωρίζετε σχετικά με τις συναντήσεις της ΑΣΕΑ ε, και των εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Των στελεχών της Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Υπάρχουν φυσικά επαφές με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας. Όπως, εμεί εμείς και εσείς έχουμε διαρκώς επαφές με όλους τους ενδιαφερόμενους. Είτε είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος, είτε με τα κράτη-μέλη, είτε με όλους. Προσπαθούμε να συλλέγουμε πληροφορίες, γιατί δεν έχουμε εμείς τη γνώση της απόλυτης αλήθειας ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσπαθούμε να συλλέγουμε στοιχεία. Οποιοδήποτε μπορεί να μας παράσχει στοιχεία, ε, τον ακούμε. Αυτό όμως δεν ε, επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις ή, λαμβάνουμε τις ε, αποφάσεις μας και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλουμε τις προτάσεις μας στο συνομοθέτη. Βεβαίως λοιπόν είχαμε επαφές και με την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. Όπως συχνά ε, συζητούμε με εκπροσώπους του, των πανεπιστημίων, των εκπροσώπων των καταναλωτών, των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων κτλ. Και τη βιομηχανία. Η συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε δεν, δεν έγινε ποτέ. Κύριε Στοζανόφσκι. I'm sorry. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποβάλω ένα ερώτημα κυρίως σε με το τι θα γίνει στο μέλλον, όχι με αυτό που έγινε στο παρελθόν, και αφορά στις ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι οποίες θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούνται από το 2017, πολύ σύντομα δηλαδή δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς ακριβώς θα γίνεται η μέτρηση, με ποιο είδους, ε, πάνω σε ποιο είδους οδηγική συμπεριφορά θα γίνεται η μέτρηση. Μήπως, για παράδειγμα, έχει συζητηθεί στην Επιτροπή, ε, στην οποία εκπροσωπούνται και τα κράτη-μέλη και τεχνικοί εμπειρογνώμονες στο ζήτημα της ε, επιβράδυνσης ή της επιτάχυνσης ξαφνικά, κάτι το οποίο είναι πολύ, εξαρτάται πολύ από τη συμπεριφορά του κάθε μεμονωμένου οδηγού. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε λοιπόν καλύτερα πώς σκοπεύουμε να γίνονται αυτές τις μετρήσεις. Λοιπόν, η οδήγηση σε, συνθήκες, ε, σε πραγματικές συνθήκες ε, είναι τμήμα, το πώς την καθορίζουμε, είναι τμήμα της όλης προσπάθειάς μας, γιατί γενικά ο τρόπος οδήγησης είναι πολύ περίπλοκος πολύ πιο περίπλοκος από το να ελέγχεις ε, σε εργαστηριακές συνθήκες ε, τις εκπομπές ενός οχήματος. Υπάρχουν δύο στοιχεία που μπορεί να προκαλέσουν αποκλήσεις. Το πρώτο είναι αυτό που θεωρούμε οριακές συνθήκες, για παράδειγμα υψόμετρο, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή θερμοκρασία και επίσης ο τρόπος οδήγησης του κάθε οδηγού. Για το θέμα του υψομέτρου, και άλλες περιβαλλοντικές συνθήκες, δηλαδή στην ουσία το γεωγραφικό σημείο που είναι το αυτοκίνητο, προβλέπουμε κάποια όρια, τα οποία είναι μέσα στους παράγοντες συμμόρφωσης και λαμβάνουν υπόψη και το ποσοστό σφάλματος, το περιθώριο σφάλματος και τις στατιστικές αβεβαιότητες. Οπότε αυτό το αντιμετωπίσαμε. Τώρα όσον αφορά τον τρόπο οδήγησης, μας ζητήθηκε να το εξετάσουμε. Αλλά θέλω να τονίσω το εξής. Θα το εξετάσουμε. Αλλά θα πρέπει να είναι ουδέτερο όσον αφορά την περιβαλλοντική επίπτωση. Η άλλη εκπρόσωπος της Κομισιόν. Κάτι ακόμη. Στο δεύτερο πακέτο RDE έχουμε βάλει τις συμπληρωματικές οριακές συνθήκες. Αυτές είναι οι παράμετροι, αυτή είναι η παράμετρος που θα μας επιτρέψει να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερα ήπια ή την ιδιαίτερα επιθετική οδήγηση. Αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ αυτών που γκαζώνουν και μεταξύ αυτών που οδηγούν σαν θίτσες. Η κυρία Μάσνα. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις είπατε ότι από το 2010 ξέρετε ότι υπάρχουν αυτές οι διατάξεις αλλίωσης, μηχανισμοί αλλίωσης. Και είπατε ότι η Κομισιόν είναι θεματοφύλαξη των συνθηκών, αυτό απαγορεύεται να υπάρχουν τέτοιε διατάξει, τέτοιοι μηχανισμοί. Και είπατε, αλλά δεν είχατε αυτέ αποδείξει ότι όντω ε, χρησιμοποιούνται τέτοιοι μηχανισμοί. Το ερώτημά μου είναι, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα πρέπει να κοιτάξετε περισσότερο. Όχι απλώ να έχετε μια ανησυχία, αλλά να ξεκινήσετε διαδικασίε παραβάση ούτως ώστε να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Και δεύτερον, και για, επειδή ξέρουμε από το 2011 τα PEMPS, έχουμε εργαστεί για αυτά, έχουμε την εντύπωση ότι χρειάστηκε πάρα πολύ μέχρι να αναπτύξετε αυτούς τους φορητούς μηχανισμούς μετρήσεων. Ανεξάρτητα από οποιασδήποτε δια, ε, διαθέσεις απάτης. Γιατί υπήρξαν αυτές οι καθυστερήσεις, για τεχνικό λόγο, τα κράτη-μέλη σας καθυστέρησαν. Γιατί έχει κρατήσει τόσο πολύ όπως ανέφερε και ο συνάδελφος Γκερμπράντι. Τα πέμπτη τα έχει από το 12 και τα χρησιμοποιεί η Σουηδία. Και εσείς ακόμη εργάζεστε γι' αυτό και είπατε το 16 στην ομάδα εργασία, γίνανε συναντήσεις για να δείτε πώς μπορείτε να τα εισαγάγετε παντού στην Ευρώπη. Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Πρώτον, εφόσον ξέραμε ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί δεν κάνετε τίποτα ή κάνατε πολύ λίγα. Και δεύτερον, γιατί τους φορητούς αυτούς τους μηχανισμούς μέτρησης όπως είπε και ο κύριος Λιούντι ακόμη δεν τους έχετε εισαγάγει με έναν τρόπο που να μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Λοιπόν, λέει της Κομισιόν, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτον, για διαδικασίες επί παραβάση των ενδεχόμενου αν θα είχαμε τέτοιο ενδεχόμενο, ε, πρέπει να καταλάβουμε οπωσδήποτε ότι είναι ένα από τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά, αλλά για να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση, πρέπει να απευθυνθεί σε ένα συγκεκριμένο κράτο μέλο. Δεν ξεκινάμε διαδικασία εν ώψη χρήση μιας τέτοιας διάταξης. η διαδικασία επί παραβάση δεν έχουμε αρμοδιότητα να την κάνουμε κατά ενό κατασκευαστή κατά μιας αυτοκινητοβιομηχανία. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαδικασία κατά ενός κράτους μέλους δεν μπορούμε να του στέλνουμε μία επιστολή. Γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη απτή απόδειξη ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνε που είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν. Αυτή είναι η διαδικασία. Και εμεί τα πορίσματα τη έρευνα τα ερμηνεύσαμε ότι δεν ήταν σε τέτοιο επίπεδο που να μα επιτρέπουν να ξεκινήσουμε διαδικασία με παραβάση. Αυτό δεν σημαίνει πω τα βρώσαμε τα χέρια. Αντίθετα, οι συνάδελφοι εξήγησαν τι έχουμε κάνει για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των υπερβολικών εκπομπών διοξιδίων αζότου. Αλλά το γεγονός ότι οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν δεν είναι κάτι που το μάθαμε τελευταία. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα με τα αυτοκίνητα. Είναι ένα ενδεχόμενο. Γι' αυτό υπάρχει νόμος που το απαγορεύει. Αλλά οποιαδήποτε στοιχεία ε, μάθαμε δεν αναφέρονταν σε συγκεκριμένη περίπτωση, σε συγκεκριμένο κράτος μέλος που θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνο. Είπατε για τα PEMS, τους φορητούς μηχανισμούς. Βεβαίως υπάρχουν πολλά PEMS, αλλά πρέπει να υποθεί ότι τα PEMS για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως χρησιμοποιούνται για ελέγχους στα βαρέα οχήματα, στα φορτηγά. Τώρα προσπαθούμε να ε, βελτιωθεί η διαδικασία για τα βαρέα οχήματα, λέει ο Μιλήτρια, των ΠΕΜΣ. Αλλά υπάρχει μια ουσιώδη διαφορά μεταξύ των μηχανισμών για τα βαρέα οχήματα, γιατί υπάρχει πολύ περισσότερο χώρο. Γιατί ξέρετε, αυτά τα ΠΕΜΣ ζυγίζουν 100 κιλά και, και των αντιστοιχών μηχανισμών για ΙΟΤΑΧΗ. Τα χρησιμοποιούμε για βαρέα οχήματα και τώρα προσπαθούμε σταδιακά να τα εισαγάγουμε και για ΙΟΤΑΧΗ. Η κυρία Μάσνερ, ναι, κάτι ακόμη για του μηχανισμού αλλίωσης. Είπατε ότι δεν είχατε καμία συγκεκριμένη υποψία αλλά είπατε ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί που είναι παράνομοι και αν έχετε ακούσει κάποιες φήμες ότι κάπου μπορεί να υπάρχουν, είχατε κάποιες ενδείξεις λοιπόν ότι κάποιος κάτι ήξερε. Γιατί δεν το ψάξατε. Κάτι ακόμη. Ήταν δύσκολο να ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση γιατί δεν υπήρχαν με βάση τον νόμο δυνατότητες επιβολής κυρώσεων. Είχε να κάνει και με αυτό. Γιατί είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι ξέρατε ότι υπάρχουν τέτοιοι μηχανισμοί που είναι παράνομοι, αλλά δεν ξέρατε που ακριβώς ήταν. Αλλά κάπου τα ακούσατε ότι υπάρχουν. Γιατί δεν το ψάξατε μετά ή δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Η ύπαρξη διατάξεων αναστολής ήταν γνωστή, αλλά δεν ήταν γνωστή η χρήση τους. Και είναι ευθύνη των κρατών μελών να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να εξασφαλίσουν ότι υπάρχει μια σωστή εποπτεία της αγοράς. Αυτό το οποίο εξήγησα συναδελφοί μου είναι ότι απουσία μια συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να ξεκινήσει η Κομισιόν διαδικασία επιπαραβάση εναντίον ενό κράτου μέλου. Χρειαζόμασταν στοιχεία. Δεν είχαμε στοιχεία. Η εφαρμογή τη νομοθεσία για την αγορά είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εμεί δεν είχαμε καμία γνώση μια περίπτωση που να χρησιμοποιήθηκαν διατάξεις αναστολής με παράνομο τρόπο στα πλαίσια της νομοθεσίας. Γι' αυτό το λόγο δεν υπήρξε καμία διαδικασία επί παραβάση. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, εγώ θα επανέλθω στο... Επειδή τέθηκε το θέμα για την ευθύνη των κρατών μελών, πρώτα πρώτα το 2013 όταν το Ερευνητικό Κέντρο προειδοποίησε για αυτά τα συστήματα αναστολής ότι μπορούσαν να αλλιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των εκπομπών. Δεν έχω καταλάβει ποια μέτρα πήρετε συγκεκριμένα. Δηλαδή, σε μια τέτοια περίπτωση ε, ε, έπρεπε να ζητήσετε συμπροματικούς ελέγχους. Και αυτό είναι το ένα μου ερώτημα. Αν ζητήθηκαν αυτοί οι συμπροματικοί ελέγχου από αυτοκινητοβιχανίες. Το δεύτερο, και ε, ποια ακριβώ ημερομηνία ενημερώσατε για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη για το πρόβλημα που εντοπίστηκε διότι δηλαδή, μέχρι σήμερα από τις ακροές αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Ενημερωθήκαμε ότι σε ένα workshop ενημερώθηκαν τα κράτη-μέλη, αλλά πότε έγινε αυτό. Το τρίτο μου ερώτημα, σήμερα ε, ενδεχομένως να υπάρχουν παρόμοια λογισμικά λύωσης και σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες, σε άλλα αυτοκίνητα πέρα αυτά από τη Volkswagen. Ε, αναφέρεστε στα κρατημέλη, αλλά να πω ότι σε ένα δημοσίευμα του Διεθνή Συμβουλίου Καθαρών Μεταφορών φαίνεται ότι παρόμοια ευρήματα των ευρώ γίνονται και στη Γαλλία σε ε, εκπομπές των αυτοκινήτων diesel και ενισχύουν την υποψία ότι αυτή η απάτη της Volkswagen δεν είναι της μόνης αυτοκινητομηχανία. Υπάρχουν και άλλες αυτοκινητομηχανίε που χρησιμοποιούν αυτά τα λογισμικά. Ε, και το ερώτημα επίσης που προκύπτει είναι κατά πόσον ε, ε, ε, έχετε εσείς πληροφορίες και στοιχεία ότι ενδεχομένως να υπάρχει αυτόν τον λογισμικό και σε άλλα αυτοκίνητα. vais répondre à la deuxième partie de votre question concernant les autres fabricants. Θα απαντήσω για το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας για τους άλλους ε, για τις άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες ενδεχομένως να εμπλέκονται. Αυτή τη στιγμή δύο κράτη-μέλη έχουν περατώσει εκθέσεις μετά από έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία. Ένα κράτος μέλος δημοσίευσε μια ενδιάμεση έκθεση η Γαλλία για τις έρευνες που συνεχίζονται. Υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη τα οποία ανακοίνωσαν θα κάνουν έρευνε και είναι εν εξελίξη. Η Κομισιόν δεν έχει πάρει καμία από αυτέ τι εκθέσει ακόμα βέβαια. Οι εκθέσει, οι οποίε είναι διαθέσιμες και η ενδιάμεση έκθεση τη Γαλλία, δηλαδή η γερμανική και η αγγλική έκθεση και η ενδιάμεση γαλλική, δεν καταδεικνύουν ότι υπήρξε παράνομη χρήση διατάξεων αναστολής από άλλους κατασκευαστές. Είπαν ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των εκπομπών στο εργαστήριο και στην πραγματικότητα. Αλλά δεν έχουν ενδείξεις για πραγματική χρήση παρα, παράνομη τέτοιων συνδικών. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμα εκφέρει γνώμη σε σχέση με τις εκθέσεις αυτές. υπάρχουν, ε, ε, υπήρξε συζήτηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της 7 η Ιουνίου. Η Επίτροπος Βιενκόφη ζήτησε από τα κράτη-μέλη να διαβιβάσουν στην Κομισιόν όλες τις πληροφορίες τεχνικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν με τις εκθέσεις αυτές και τις αναλύσεις που περιέχονται σε αυτές. Γιατί χωρίς αυτές τις πληροφορίες δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε τις εκθέσεις και τα συμπεράσματα των κρατών μελών για αυτά τα θέματα. Αυτή τη στιγμή οι εκθέσεις αυτές αφορούν τα οποία κάνουν ερεύνες, όχι για την, για την παράνομη αυτή η χρήση. Η Κομισιόν όμως δεν είναι σε θέση να εκφέρει γνώμη αν δεν έχουμε τις λεπτομεριακές πληροφορίες από τα κρατη και επίσης τις πληροφορίες που θα έρθουν από εκθέσεις άλλων χωρών. Δεν μπορούμε εμείς να ε, εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε τις εκθέσεις αυτές χωρίς τα στοιχεία αυτά. Για το πρώτο τμήμα της ερώτησής σας, για την έκθεση του 2013, ρωτήσατε αν τα κράτη-μέλη ήταν ενήμερα για τα πορίσματα της έρευνας από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η απάντηση είναι ναι. Η, έρευνα, η έκθεση του Κοινού Κέντρου Έρευνας ήταν μια δημόσια έκθεση και παρακολουθήθηκε από όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών και τις αρμόδιες αρχές επιοπτείας της αγοράς. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι η έκθεση του 2013 αφορά μια σειρά από εργασίες που είχαν σαν στόχο να επιτευχθεί μια ε, μέθοδος αξιόπιστη και ανθεκτική η οποία μπορούσε να οδηγήσει σε μέτρηση των πραγματικών εκπομπών. Θα ήταν καινοτόμα αυτή η μέθοδος γιατί με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιούνται διατάξεις αναστολής ώστε τα προβλήματα του παρελθόντος να μην μπορούν να επαναληφθούν. Ε, γιατί ήταν στο παρελθόν μεν τα συστήματα αυτά αλλά δεν μπορούσαν να ανοιχνευτούν. Και ο εκπρόσωπος του Κέντρου Ερευνών τόνισε ότι υπήρχαν καινοτόμα στοιχεία στην ε, πρόταση αυτή για να μην μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές αναστολής. Αν έγινε κατάλληλη προσπάθεια να φέρουμε στην προσοχή των κρατών μελών το θέμα του σεβασμού των κοινοτικών κανόνων για τις εκπομπές από τα οχήματα. Βεβαίως το κάναμε αυτό. Τονίσαμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο η εποπτεία της αγοράς. Αυτό συζητήθηκε και με τρόπο αρκετά διάφανο στην ε, ομάδα εργασίας για τα οχήματα, όπου εμείς πιέσαμε να υπάρξει περαιτέρω αναστοχασμός για τον κατάλληλο χαρακτήρα των εργαλείων που έχουμε για την εποπτεία της αγοράς. Αυτές οι αναστοχαστικές συζητήσεις οδήγησαν σε μια τροποποίηση του κανονισμού που ε, ενεκρίθη τον Ιανουάριο του 2016 με πρόταση της Επιτρόπου Μπιανκόφσκα. Το 2016 ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα βιομηχανίας έστειλε μια επιστολή στα κρατη για να τους ζητήσουν να παρακολουθήσουν εναργώς και με μεγάλη προσοχή τις, ε, τους κανονισμούς για την ε, εποπτεία της αγοράς για να μην αποδυναμωθούν οι κανόνες σε σχέση με την ασφάλεια και την λειτουργία της αγοράς. Αυτό έγινε το 2013 μαζί με τις ε, Προ πρόοδου στο θέμα των ε, πραγματικών εκπομπών, των δοκιμασιών πραγματικών εκπομπών. Κύριε Σιλικιώτη ήδη έχετε μιλήσει για 7 λεπτά, θα επανέλθουμε. Θα έπρεπε να ζητήσω από του εκπροσώπου τη Κομισιόν να είναι πιο επακριβεί σε αυτά που λένε και να μην επεκτείνονται σε εξηγήσει οι οποίε είναι παράπλευρε για τα θέματα αυτά. Κύριε Σιλικιώτη, πάρα πολύ σύντομα είναι εδώ ότι ενώ μιλούμε για τις ευθύνε των κρατών μελών, ενώ ακόμα και στις γραπτές ε, απαντήσεις που μας στείλατε, το ερώτημα που προκύπτει είναι η δική σας η ομάδα είναι υπεύθυνη να παρακολουθά την ανάπτυξη των πολιτικών των κρατών μελών και να διασφαλίζει την εφαρμογή τη σαν νομοθεσία. Και το ερώτημα είναι ακριβώ τι έχετε κάνει για να επισπεύσετε. Δεν αρκεί κύριε Κοζούκου να λέμε ότι αναμένουμε εκθέσει από τα κρατη Ε, πρέπει και εσεί να ενεργήσετε σε επιτροπή απέναντι στα κρατη Okay. Είναι το θέμα των εθνών σας, ναι ή όχι αυτό. Ναι, χωρίς να μακρηγορήσω, είναι α, μέρος των υποχρεώσεών μας και κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο για να τις ατηρήσουμε αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποστηρίξει της πρωτοβουλίες από την Κομισιόν όταν διαπιστώθηκε για παράδειγμα ότι ένας κατασκευαστής δεν τηρούσε τις προδιαγραφές για τον κλιματισμό. Ε, τότε ανέλαβε πρωτοβουλία σχετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριο Σέκχαρτ, είναι απογοητευτική αυτή η ανταλλαγή, γιατί δεν μας δίνεται συγκεκριμένες απαντήσεις. Και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Στην γραπτή μας ερώτηση, ρωτήσαμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνώριζε ότι υπήρχαν ε, συστήματα μέτρησης της θερμοκρασία έτσι ώστε να μειώνονται οι εκπομπές κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μας απαντάτε όχι. Όμως υπάρχουν έγγραφα και η απάντησή σας τώρα μόλις ε, μας είπατε ότι το JRC γνώριζε ότι διατάξεις χρησιμοποιούνται για την ε, αλλίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε χαμηλέ θερμοκρασίε. Αυτό το 2013. Επομένω είναι στοιχεία τα οποία ήταν αναπολύτω γνωστά από το 2013. Ενώ στην γραπτή σα απάντηση μας λέτε δεν το γνώριζαμε. Αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ένα ψέμα. Επίσης μας λέτε ότι τα συστήματα αυτά αφορούν, ε, Μα είπατε εσεί μόλι τώρα ότι τα συστήματα αυτά αφορούσαν διζολοκίνητα αυτοκίνητα. Επομένω, μην μα δίνετε ψεύτικε πληροφορίε. Πώ είναι δυνατόν στην γραπτή σα απάντηση να μα λέτε ότι δεν το γνωρίζετε, όταν εδώ έρχεστε και μα λέτε ότι υπάρχουν τέτοια λογισμικά. Και ο κ. Ε, Φάλκενμπερ μα λέει ε, ότι υπάρχουν τέτοιε τεχνικέ. Θα ήθελα να λάβουμε μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό, λέει η Πρόεδρος. Δώσαμε πολύ χρόνο σε όλους, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ κρίσιμη η διαφορά μεταξύ αυτού που αναφέρεται στην επιστολή του κ. Φάλκενμπεργκ και των απαντήσεων που μας έδωσε η Επιτροπή στις γραπτές ερωτήσεις της. Στις γραπτές μας ερωτήσεις. Δεν εθιμούμε αλλά την εποχή εκείνη οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν εστιάσει στην ανάπτυξη των μηχανισμών μέτρησης της πραγματικής συνθήκης, το RDE. Αυτή ήταν η πρώτη οριότητα. Για να έχουμε μια μέτρηση που να λειτουργεί σωστά. αναφέρεται, αυτό που αναφέρεται, ε, είναι μία... Μάλλον, δεν υπάρχει συγκεκριμένο στοιχείο. Παρέμβαση. Όμως, στη συνέχεια της επιστολής ζητείται από την TG Enterprise να εξετάσει την νομιμότητα, να διερευνήσει μάλλον την νομιμότητα της χρήσης τέτοιων παρακτικών. Όμως, την απάντηση της Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας δεν απάντησε σε αυτό. Επομένως, αυτό που συζητάμε είναι ότι σας ζητήθηκε να διενεργήσετε μια έρευνα και να το πράξατε. Απάντηση τη Επιτροπή. Η προτεραιότητά μας τότε ήταν να ε, ε, αναπτύξουμε τη διαδικασία αυτή e και όπως σας είπα και πριν χρειαζόμασταν αποδεικτικά στοιχεία. Παρέμβαση. Γι' αυτό ζητήθηκε να διενεργηθεί έρευνα. Εάν είχατε διεξάγει την έρευνα, θα είχατε τα στοιχεία που σας χρειαζόντουσαν. Η πρόεδρος μας έδωσαν την απάντησή τους, δεν ήταν προτεραιότητα, η προτεραιότητα τους ήταν το RD. Το μέλος της Επιτροπής, ε, ναι, αλλά τότε να μας απαντήσετε έτσι, να μας πείτε δεν ήταν προτεραιότητα. Δεν το βρήκατε γιατί δεν το ψάξατε. Επειδή μου λένε να είμαστε επακριβείς, θα προσπαθήσω να είμαι επακριβής. Η Guardian αναφέρεται σε λαθασμένα συνέχεια Μα μου ζητήσατε να υπάρχει μία εξήγηση. Εγώ έδωσα την εξήγηση μου γιατί ήταν το ερώτημα που είχε να κάνει με το άρθρο του Guardian. Το άρθρο του Guardian αναφέρεται στα πρακτικά και εγώ εξήγησα ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την, με την επιστολή Φάλκεμπεργκ. Εντάξει, θέλετε να είμαστε επακριβείς. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε την απάντησή σας στο ερώτημα υπαριθμό 8. Ένα άλλο παράδειγμα ότι όχι μόνο δεν είσαστε ακριβείς στις απαντήσεις σας, αλλά δεν φαίνεται να καταλαβαίνετε τι λέει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νομοθεσία λέει ότι ο κατασκευαστής θα εξοπλίσει τα οχήματα έτσι, ώστε τα τμήματα της, του κινητήρα που μπορούν να επηρεάσουν τις εκπομπές θα εξασφαλίσουν ότι το όχημα σε φυσιολογικές συνθήκες θα συμμορφώνεται με τον κανονισμό. Αυτό είναι το άρθρο 5 του κανονισμού γύρω 6. Επομένως τα αυτοκίνητα πρέπει να συμμορφώνονται κατά τη διάρκεια φυσιολογικής χρήσης. Και έρχομαι τώρα στην απάντησή σας στο ερώτημά μας 8. Λέτε, εφόσον το σύστημα έγκρισης τύπου εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη και συμμορφώνεται με τα ε, όρια α, ε, οξυδίων αζότου στο εργαστήριο. Όχι, ο μόνος λέει ότι πρέπει να συμμορφώνται σε πραγματικές συνθήκες. Που λέει, νόμος που λέει η νομοθεσία ότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση σε συνθήκες εργαστήριου. Δεν το λέει πουθενά. Εσείς λοιπόν για ποιο λόγο έχετε αλλάξει το γράμμα του νόμου και λέτε ότι μόνο στο, εργοστάσιο, στο, εργοστάσιο, στο εργαστήριο πρέπει να <clears throat> υπάρχει συμμόρφωση στην έγγραφη απάντησή σας προς την Επιτροπή μας. Sure, I answer your question. Just... Βεβαίως, θα απαντήσω. Όπως σωστά λέτε, ο κανονισμός του 2007 7-15 αναφέρεται σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Ωστόσο, τα όρια ορίζονται για μια συγκεκριμένη διαδικασία τεστ, γιατί ο κανονισμός ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει και να εισαγάγει διαδικασίες ελέγχου, διαδικασίες τεστ. Η Επιτροπή λοιπόν εισήγαγε διαδικασίες για τη μέτρηση των καυσαερίων και οι διαδικασίες οι προηγούμενες ε, ήταν πάντα εργαστηριακές. Έχετε δίκιο. Μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι ιδανικές ε, οι συνθήκες για ένα τεστ εργαστήριο και εφόσον συμμορφούνται μόνο σε εργαστήριο με κάποιες οριακές τιμές, τότε δεν εφαρμόζεται πλήρως ο νόμο. Αλλά δεν μπορείτε να στραφείτε κατά ενός κατασκευαστή ή κατά μιας ρυθμιστικής αρχής, εφόσον συμμορφούνται με τις διαδικασίες. Ε, έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε διαδικασίε, αλλά στο παρελθόν οι διαδικασίε που είχαμε, οι δεσμευτικέ, ήταν εργαστηριακές για να μετρήσουμε και τα οξύδια του αζότου και άλλα. Τώρα αλλάξαμε γιατί θεωρώ το άρθρο 14 μας δίνει τη δυνατότητα ή καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή δίνει εντολή στην Επιτροπή να εισαγάγει αυτές τις νέες διαδικασίες και, τις, και εισήχθησαν. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούσαν τις διαδικασίες τεστ που είχαν ήδη εγκριθεί, ανάλογα με την υπάρχουσα εντολή και αρμοδιότητες. Ο κύριος Έκουτ, να καταλήξω. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τα άτομα αυτά, αλλά μόνο μετά που θα έχουμε δει όλη την ανταλλαγή email με το κοινό κέντρο ελέγχου και με άλλους σημαντικούς φορείς. Μόνο άμα δούμε όλοι σας την επικοινωνία θα <clears throat> μπορούμε να κάνουμε ουσιαστική συζήτηση. Πρόεδρος, ναι, θα το συζητήσουμε με τους συντονιστές γιατί θα πρέπει να δούμε και τις πολιτικές ευθύνες. Ο κύριος Τζούλο. Είμαι λιγάκι μπερδεμένος με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα <clears throat> σε αυτή την ε, συζήτηση είναι σαν να ζούμε σε δύο παράλληλους κόσμους. Εσείς λέτε για προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι προτεραιότητες, για κανονισμούς οι οποίοι δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά τι γίνεται. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Πράγματι ισχύουν αυτά τα οποία βλέπουν. Ε, λέτε ότι δεν είχατε καθόλου στοιχεία <clears throat> για την ύπαρξη συσκευών διατάξεων ε, αναστολής. Αλλά σήμερα, όχι μόνο εγώ, όχι συναδελφοί μου έχουμε κάπως ε, ανακατασκευάσει το ιστορικό με την ε, επιστολή αυτή που είχε να κάνει με τις, ε, με έρευνες που έγιναν στο κέντρο ερευνών που έδειχνε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες ε, ατασταλίες στα θέματα αυτά. Επίσης, έχουμε την επιστολή από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος η οποία προειδοποιεί ότι υπάρχουν παράνομες ε, διαδικασίες. Έχουμε την αλληλογραφία του Νοεμβρίου του 2014 πάλι μεταξύ του κυρίου Φάλκεμπερ και του Γενικού Διευθυντή του, τμήμα, του, της ε, Υπηρεσίας Βιομηχανίας στην Κομισιόν. Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι δεν υπάρχουν καθόλου ενδείξεις. Αυτό είναι ανησυχητικό. Ήταν απαραίτητο να ερευνήσετε περισσότερο, εσείς όμως προτιμήσατε να δώσετε προτεραιότητα σε κάτι άλλο γιατί δίνεται πιο μεγάλη σημασία στις διαδικασίες από ότι στην επίλυση των προβλημάτων. Ακόμα και από τις σημερινέ απαντήσεις έχουν έλθει στην επιφάνεια κάποια στοιχεία που είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Υπάρχει το πρόβλημα λοιπόν με τη μέτρηση των ε, εκπομπών σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας. Αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί στο μέτρο. Λέτε ότι δεν έχετε δεδομένα συγκεκριμένα στοιχεία και θα πρέπει δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Λοιπόν, πού πρέπει να, τι σύστημα είναι αυτό στο οποίο περιμένετε πρώτα να έρθουν τα πράγματα στο φως και όχι να προσπαθήσετε να προλάβετε τις ε, απάτες. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να καταλάβουμε αν και πότε η Κομισιόν πίεσε τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Σας ζητώ λοιπόν να αλλάξετε την προσέγγισή σας και να είσαστε πιο τίμοι, πιο ειλικρινείς ενώπιον της Επιτροπής μας, ώστε να μπορέσει η πραγματική προβληματική αυτή να προχωρήσει και να ξεπεράσουμε τα σκάνδαλα αυτά τα οποία είδαμε. Θέλω τώρα να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τις συσκευές φορητής ε, καταμέτρησης ε, εκπομπών, PEMS. Λέτε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένας παράγον συμμόρφωσης για να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες ε, περιβαλλοντικές οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη μέτρηση με τα PEMS αλλά οι κατασκευαστές αυτών των συσκευών λένε ότι η αβεβαιότητα δεν ξεπερνάει το 20 με 30% και ενδεχομένως στο μέλλον θα είναι μονάχα 15%. Γιατί λοιπόν αυτή η τόσο χαμηλή αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την μέτρηση οδηγεί σε ένα παράγοντα συμμόρφωσης ο οποίος πρέπει να είναι πολύ ψηλότερο από αυτό που χρειάζεται για να καλύψει την αβεβαιότητα της ε, ε μέτρησης. Από τι άλλο εξαρτώνται λοιπόν αυτοί οι παράγοντες συμμόρφωσης, αν δεν είναι μονάχα η αβεβαιότητα των μετρήσεων. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σχολιάσω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε να δώσουμε έντιμες και ειλικρινείς απαντήσεις. Δεν πρέπει να μας κατηγορείτε ότι δεν είμαστε ειλικρινείς ενώπιον της εκτροπής. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα. Νομίζω ότι εξηγήθηκε στην προηγούμενη ακρόασή σας με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ε, ελέγχθη σαφώς ότι ο εξοπλισμός PEMS για τα επιβατικά οχήματα πρέπει να πλησιάσει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στα βαρέα επαγγελματικά ε, οχήματα, βελτιώνεται, αλλά αν έχει χρησιμοποιηθεί για πολλές ώρες η βαθμονόμηση του εξοπλισμού μπορεί να αλλάξει. <clears throat> Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε αυτές τις λεπτομέρειες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν περαιτέρω για να μειωθεί η αβεβαιότητα της μέτρησης, την οποία αναφέρεται και εσείς ο ίδιος. Ε, Εντάξει, λοιπόν, αυτό το όριο όμως το οποίο έχετε εσείς θέσει, το όριο αβεβαιότητος, δεν έχει να κάνει με τις ε, μελέτες, κάπως το έχετε βγάλει από ένα καπέλο εσείς. Δεν στοιχειο, δεν στοιχειοθετείται <clears throat> από τον τωρινό εξοπλισμό. Γιατί πρέπει να έχετε μια, <clears throat> ένα περιθώριο αβεβαιότητας 80% αν δεν είναι αυτή η αβεβαιότητα των τωρινών μετρήσεων. Ευχαριστώ. Υπάρχει πράγματι η αβεβαιότητα στις μετρήσεις ΠΕΜΣ <clears throat> και νομίζω ότι είπαμε ότι εξετάζουμε σε εργαστήριο τις ε, ε αβεβαιότητες αυτές γίνεται ε, έλεγχος σε εργαστηριακό επίπεδο και αυτό μας δίνει περίπου το 30% βεβαιότητας που λέτε. Αλλά αυτό το αποτέλεσμα συζητήθηκε στην ομάδα RDLTV, την ομάδα εργασία για τα ελαφρά οχήματα και υπήρξαν περαιτέρω σχόλια, περαιτέρω αναλύσεις και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι αν μετράτε το, στο εργαστήριο και μετά βγείτε από το εργαστήριο θα αυξηθούν οι αβεβαιότητες. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρθηκε αυτή η αβεβαιότητα της τάξης του 50% αλλά υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης που θεωρεί ότι εάν βελτιωθεί η ακρίβεια των συσκευών θα μειωθεί η αβεβαιότητα. Για το συγκεκριμένο σας ερώτημα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία τύπου, έγκρισης τύπου και τα PEMS, αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο και εμείς το αποδεχόμαστε και αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι συσκευές PEMS μπορούν να πιστοποιούνται και να εγκρίνονται με έναν τρόπο ο οποίος θα οδηγεί σε ομοιογενή αποτελέσματα σε όλες τις συνθήκες χρήσης. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε κλείσει τον πρώτο γύρο. Νομίζω ότι έδωσα σε όλους λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι απαντήσεις που θέλουμε να πάρουμε και δεν είναι θέμα χρόνου. Πρέπει όμως να τελειώσουμε καιρός και πρέπει να υπάρχει ισότης ευκαιριών για όλους τους ομιλητές τη Επιτροπή μα. Παρακαλώ λοιπόν παραμείνετε στο χρόνο που αναφέρεται. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο γύρο με πέντε λεπτά για τους εισηγητέ και του εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ παραμείνετε στα χρονικά όρια, σύντομε και περιεκτικές ε, ερωτήσεις και παρακαλώ να είναι και οι απαντήσεις ανάλογα συγκεντρωμένες και συνοπτικές. Ευχαριστώ. Επανήλθα. Παρακολουθώ λοιπόν αυτή τη συζήτηση και συμφωνώ με αυτά που είπαν συναδελφοί ότι δεν είναι μονάχα το θέμα των διατάξεων αναστολής. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Είδαμε τι γίνεται με τις τράπεζες, με, τα, με τις δοκιμασίες αντοχής, ότι δοκιμάζουμε σε διάφορες συνθήκες. Είναι σαν να δοκιμάζει κανείς σε διαφορετικές συνθήκες, αλλά και για τις εκπομπές των οχημάτων. Εξακολουθώ να διαβάζω, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είχα διαβάσει προηγουμένως και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον. Τα πορίσματα του εργαστηρίου σας το 2010. Σελίδα 6. Καταλήγει στο ότι, ότι χρειάζεται μια ομάδα για τις δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες με προσώπους των κρατών μελών και της βιομηχανία. Το 2010 το λέει αυτό η Κομισιόν, ώστε να παρακολουθήσει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δοκιμασίας RDE για τα οχήματα Euro 6. Και μετά λέτε ότι η μέθοδος αυτή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη στο τέλος του 2012 για να εγκριθεί με διαδικασία επιτροπολογίας. Η ομάδα RDE θα πρέπει να συνεδριάσει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2011. Εδώ και πολλά πολλά χρόνια λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο κατάλαβε ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία μεταξύ εκπομπών οξυδίου του αζότου και διοξυδίου του άνθρακος, αλλά και ότι οι πραγματικές μετρήσεις δεν πρέπει να γίνονται στο εργαστήριο, αλλά σε πραγματικές συνθήκες, όπως γίνεται και με την ανθρώπινη καρδιά, όχι μονάχα στο ιατρείο, αλλά και σε πραγματικές συνθήκες. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητήσω την ικανότητα των τεσσάρων σας ή την ικανότητα της Κομισιόν. Νομίζω ότι είσαστε ιδιαίτερα ικανοί άνθρωποι. Το ερώτημά μου είναι όμως τι έγινε, ποιος τροχοπέδησε αυτή τη διαδικασία, γιατί σταμάτησε αυτή η διαδικασία, γιατί δεν κάνατε αυτό το οποίο προβλέπατε να κάνετε. δεν σταμάτησαν οι εργασίε. Μπορώ να σα δώσω πολλά στοιχεία που μπορούν να σα βοηθήσουν να καταλάβετε τι ακριβώ έγινε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία εξέβρεση μιας αξιόπιστης μεθόδου. Αυτό έγινε κατά τα έτη 2012, 2013, 2014. Χρειάστηκε να αξιολογήσουμε όλες τις πληροφορίες που είχαμε και ναι, καταλαβαίνω Στοιχεία, στοιχεία, στοιχεία που πρέπει να αξιολογήσετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο κύριο Κάρνη. Εσείς οι ίδιοι όμως είπατε ότι η μέθοδος αυτή θα πρέπει να είναι έτοιμη στο τέλος του 2012. Το 2010 φαίνεται ότι είχατε αρκετά στοιχεία ώστε να καθορίσετε, ξέρετε που είναι το πρόβλημα και το ξέρετε πολύ καλά. Φαίνεται λοιπόν ότι ξέρετε πόσο χρειάζεται να εργαστείτε για να καταλήξετε. Είναι τόσο βαριά και επαχθή σε αυτή η διαδικασία ώστε από το 2010 στο 2017 είναι μια ταχεία διαδικασία ενώ λέγατε το 2012 ή υπάρχουν κάποια άτομα και κάτι μέλη που παρενέβησαν, είπανε, σε καμία περίπτωση πάνω από το πτώμα μας, το ξέραν αυτό οι επίτροποι, το ξέρανε τα μέλη της Κομισιόν. Κάποιος φαίνεται ότι απλώς εμπόδιζε όλη αυτή τη διαδικασία και ποιος το έκανε. Για δύο λόγους καθυστερήσανε ε, αυτές οι εργασίε Κατά τη διάρκεια του 2012-2013 υπήρχαν τεχνικές δυσκολίες στο να καταλήγουμε ποια θα ήταν η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος. Στην έκθεση του 2013 του Κοινού Κέντρου Έρευνα υπάρχει μια πολύ αναλυτική καταγραφή όλων των βημάτων που έγιναν έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλες οι τεχνικές μέθοδοι που ήταν διαθέσιμες για να καταλήξουμε σε μια ε, διαδικασία μέτρησης των εκπομπών πιο αξιόπιστη από εκείνη που είχαμε ε, με την εργαστηριακή μέτρηση. Μετά θα έπρεπε να βρεθεί στην Επιτροπή TCMV η συμφωνία με τα κράτη-μέλη. Αυτό μας καθυστέρησε κατά τη διάρκεια του 2014 γιατί απεδείχθη ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι περιμέναμε ε, να υπάρξει υποστήριξη και η η η ειδική πλειοψηφία το 2014. Τώρα καταλάβαμε, λέει ο μιλητή, ποιο ήταν εκείνο που καθυστερούσε το 2014. Απάντηση τη Επιτροπή. Δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι εδώ ε, χρειάζεται ειδική πλειοψηφία, άρα να υποστηρίζουν την πρόταση ένα μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Ερώτηση. Και ποιε ήταν ακριβώ αυτά τα κράτη-μέλη που δεν υποστήριζαν. Απάντηση τη Επιτροπή. Ε, τρεις, σε τρεις κατηγορίες θα μπορούσα να ε, τα κράτη-μέλη. Υπήρχαν κάποια κράτη-μέλη τα οποία υποστήριζαν ένθερμα και τα οποία θα ήθελαν αυτή η διαδικασία να προχωρήσει γρήγορα. Για παράδειγμα η Δανία ή η Ολλανδία. Δεύτερη κατηγορία είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες επιθυμούσαν μια προσεκτική διαδικασία έτσι ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους κατασκευαστές να ε, προσαρμοστούν. Αυτά τα κρατημέλη ήταν κυρίως του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης. Το θέμα συζητήθηκε διαρκώς και ενδελεχώς στην TCMV. Προσπαθούσαμε να καταλήξουμε σε συμφωνία, σε συνένεση και τελικά η ψηφοφορία έγινε στις 19 Μαΐου του 2015. ευχαριστώ. Δυσκολεύομαι να καταλάβω το εξής. Σήμερα είμαστε ικανοί να μετρήσουμε τα οξύδια του αζότου στον Άρη. Και ταυτόχρονα μας λέτε ότι χρειαζόμαστε χρόνια, χρόνια, πολλά χρόνια για να καταλήξουμε σε μία ε, μεθοδολογία μέτρησης των οξυδίων του αζότου που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα, τα οποία είναι ε, δισεκατομμύρια στον πλανήτη μας. Ε, δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς τα μετράμε τόσο εύκολα στον Άρη και τόσο δύσκολο στη Γη. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε, ότι, είναι ότι υπήρχε δυσκολία στην, στο να βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία που χρειαζόταν. Αυτό σημαίνει όμω ότι υπήρχαν κράτη-μέλη που μπλόκαραν τη διαδικασία και θα ήθελα να τα ονοματίσετε αυτά. Ποια ήταν ακριβώ τα κράτη-μέλη που καθυστερούσαν τη διαδικασία. Επίση, αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι δύσκολο τεχνικά να βρεθεί μια μέθοδο για να μειωθούν οι εκπομπέ. Αυτό ναι. Αλλά αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι είναι γιατί είναι δύσκολο να βρεθεί μια μέθοδο μέτρηση. Απάντηση τη Επιτροπή. υπήρχαν κράτη-μέλη τα οποία δεν συμφωνούσαν με τη διαδικασία ή με τα όρια, αλλά το γεγονό ότι δεν συμφωνούσαν με τα όρια ή με τη διαδικασία δεν σημαίνει ότι μπλόκαραν. Ναι, εγώ δεν σας ρωτώ για πέρυσι, σας ρωτώ για το 2011-2012. Τι συνέβαινε τότε, ποια ήταν ακριβώς εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία εμπόδιζαν τις εξελίξεις και κολλησιεργούσαν. Είναι κάτι το οποίο ανέφερα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, της προάλλες. Ένα παιδί 8 χρονών καταλαβαίνει ότι για να μετρήσεις τι εκπέμπει ένα αυτοκίνητο πρέπει να το μετρήσεις στην εξάτμιση. Και χρειάστηκαν χρόνια επί χρόνων για να το αντιληφθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί. Για το 2012-2013 οι συζητήσει που γινόντουσαν ήταν κυρίω τεχνικού χαρακτήρα στο επίπεδο τη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και τι λεπτομέρειε αυτών των συζητήσεων, το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων μπορείτε να τι βρείτε στην έκθεση του Κοινού Κέντρου ε, Έρευνα. Ε, δεν υπήρχε μια συγκεκριμένη πρόταση επιτάπητο. Αυτό που συζητούσαμε ήταν η παράμετροι και η μεθοδολογία. Εκείνη την εποχή, από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, ήλπιζε ότι δεν θα χρειαζόταν τόσο πολύ χρόνο, τελικά χρειάστηκε περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια μεθοδολογία που είναι τελικά αυτή η μεθοδολογία που ε, κατέγραψε στην πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μετά συζητήθηκε με τα κράτη-μέλη ο μεταβατικός χρόνος ε, που θα χρειαζόταν, ο χρόνο που θα χρειαζόταν για να τεθούν αυτά τα πράγματα σε εφαρμογή και αυτό συζητήθηκε κατόπιν όλη τη διάρκεια του 2014. Ερώτηση. Ναι, με όλα αυτά που μου λέτε, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώ βρισκόταν και δεν είχε μια ενεργό συμμετοχή. Εσεί γιατί το επιτρέψατε αυτό, γιατί επιτρέψατε να κολλησιεργούν τα κράτη-μέλη και γιατί επιτρέψατε να χρονίζει αυτή η συζήτηση για τα τεχνικά θέματα. Αυτή η εικόνα που δείχνει σήμερα το πρωί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι εμείς απλώς προεδρεύαμε. Είμαστε εκεί, αλλά τα κράτη-μέλη. Επανέρχομαι στη γραπτή ερώτηση 7. Αναφέρεται ότι στον κανονισμο 7.15.2007 δεν προβλέπεται ρητά ότι ο, ο, ο κατασκευαστής οφείλει να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την, ε, της, την εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρου 5.2 για τις διατάξεις αναστολής. Ωστόσο, ο κανονισμός αναφέρει ότι θα πρέπει να παρέχει ο κατασκευαστής πληροφορίες για το σύστημα ανακύκλωσης καυσίμων συμπεριλαμβανομένης και της συμπεριφοράς του σε χαμηλές θερμοκρασίες. Καυσαερίων. Ανακύκλωση Γιατί λοιπόν ποτέ δεν χρησιμοποίησατε αυτόν τον κανονισμό του 2008 για να σας δώσουν ε, οι κατασκευαστές μέσω των κρατών μελών τις σχετικές πληροφορίες για να διευκρινίσουν πώς χρησιμοποιούν ε, και αν χρησιμοποιούν διατάξεις αναστολής. Ή τουλάχιστον να εξηγήσουν ε, πότε χρησιμοποιούν και πότε σταματά το αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους μείωσης των εκπομπών του. Ναι. Υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ της υποχρέωσης που αναφέρατε και που τώρα είναι τμήμα της διαδικασίας RDE2 είναι η δήλωση που κάνει ο κατασκευαστής. Ναι, αυτό το, το εισάγαμε για να ε, υποχρεώσουμε τον κατασκευαστή να κάνει κάτι που εκπεφρασμένα δεν προβλεπόταν από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή την ερώτηση θα την απαντούσαν καλύτερα οι αρχές έγκρισης τύπου, γιατί αυτοί πρέπει να ελέγξουν αυτές τις πληροφορίες. Ο κατασκευαστής πρέπει να δώσει στην αρχή έγκρισης τύπου τα στοιχεία για τα συστήματα προστασίας των κινητήρων και η εθνική αρχή πρέπει να ελέγξει. Άρα ε, οι πιο ενδεδειγμένοι για να σα πω αν το έκανα, είναι οι αρχέ έγκρισης τύπου των κρατών μελών. Αλλά, επιπλέον, Τώρα με το δεύτερο πακέτο RDE ζητάμε συγκεκριμένα από τους κατασκευαστείς να μας πούνε ποιες είναι οι βασικές και οι επιπλέον εκπομπές. Ναι, λέει ο κύριος Γκέμπραντι, αλλά αυτές είναι ο κανονισμός του 2008. Τόσα χρόνια. Εσείς μου λέτε να ρωτήσω τις αρχές έγκρισης τύπου, γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν γνωρίζουμε πώς εφαρμόζεται αυτός ο κανονισμός. Η Επιτροπή αυτό που είπα είναι ότι υπάρχει μια αλυσίδα ευθυνών. Η έγκριση τύπου, επειδή το σύστημα είναι συγκεντρωτικό, είναι τα κράτη-μέλη που εγκρίνουν τα αυτοκίνητα. Αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν τι προφορίε που παρέχουν οι κατασκευαστέ. Ευχαριστώ κύριο Κάρεν. Να μιλήσω ο κύριο Γκίζη κάτι για μένα. Ε, να ξεκουραστεί λίγο ο συνάδελφο Κάρεν. Έχει κάνει τόσε καλέ ερωτήσει. Εγώ ε, ω του ΕΛΚ ε, είμαι στην ε, περίεργη θέση ότι συμφωνώ με τον συνάλφο Έιχοτ Διότι αυτά που ακούμε είναι λίγο ανισχυτικά και η πληροφόρηση που λαμβάνουμε δεν είναι πολύ συγκεκριμένη. Να δούμε χρονολογικά πώ μπορώ να συνοψίσω την κατάσταση. Διαπιστώσαμε, κύριε Κοζιγκού, ότι από το 2007 γνωρίζουμε ότι οι εκπομπέ αζότου των διζελοκινητήρων είναι υψηλέ. Και στα πλαίσια της διαδικασίας επιτροπολογίες που βέβαια ο απλός πολίτης δεν ξέρει τι σημαίνει. Δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα εργασίας για τα οχήματα από το 2011 και καταλήγουμε σε ένα νόμο RDE για να λύσουμε το πρόβλημα το 2015 όπου θα γίνει ακόμη πιο αυστηρή νομοθεσία το 17. Δηλαδή, 7 ξεκινήσαμε, 17 καταλήξαμε. Μια δεκαετία. Εάν παρατηρούσατε απ' έξω τη διαδικασία, Πώς θα εκτιμούσατε. Τι βαθμό θα τις βάζετε. Ε, λέει ο πρόσωπος Κομισιόν. Καταρχάς, καταρχάς, να διευκρινίσω τις πληροφορίες που σας έχουμε ήδη δώσει για να υπάρχει η ίδια κατανόηση. Είναι γνωστό ότι τα οξύδια του αζότου είναι πρόβλημα και δεν ξεκίνησε η προσπάθεια ελέγχου του στο 2013 ελέγχονται από την προϋπάρχουσα νομοθεσία, εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή για τις εκπομπές αυτές. Το πρόβλημα όμως είναι ότι τα τεστ που χρησιμοποιούσαμε δεν ανταποκρίνονταν στις πραγματικές εκπομπές. Και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο εντοπίσαμε. Και όταν το εντοπίσαμε, ξεκινήσαμε να προσπαθούμε να το επιλύσουμε, αλλά ήταν περίπλοκη τεχνική η διαδικασία, κράτησε περισσότερο από ό,τι όλοι θα θέλαμε και θα ελπίζαμε αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα τεστ που να μετράει τις πραγματικές εκπομπές. αυτό κάναμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέραμε ότι υπάρχουν οξύδια του αζότου, ξέραμε τις επιπτώσεις τους, ξέραμε ότι ήταν επιβλαβή και ότι δεν κάναμε τίποτα για όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Ξέραμε για το οξύδιο του αζότου, υπήρχε νομοθεσία, Ξέραμε για τον κίνδυνο μηχανισμών αλλίωσης, απαγορεύονταν. Υπήρχε ένα θέμα με τα τεστ που είχαμε εφαρμόσει γιατί ήταν ανεπαρκή. Και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε τα τεστ. Να σας διακόψω. Δεν είπατε κάνετε τίποτα. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Κάτι κάνατε, αλλά δεν συμφωνείτε ότι 10 χρόνια από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε το πρόβλημα μέχρι να υπάρξει νομοθετική αντιμετώπιση του τα είχαμε παλιά στα κομμουνιστικά καθεστώτα, ότι είχαν δεκαετή πλάνα. Έτσι λοιπόν λειτουργεί και η Κομισιόν. Um, allow to... Επιτρέψτε να κάνω ένα σχόλιο ως κάποιος που βρίσκεται ως κάποιος που δεν είναι πια υπάλληλος της Κομισιόν βρίσκομαι έξω από αυτή τη διαδικασία, δεν έχω ασχοληθεί με την νομοθεσία τα τελευταία δέκα χρόνια. Είμαι ένας εξωτερικός παρατηρητής, αν θέλετε. Όταν ήμουν επικεφαλής της ομάδος για τα, μονάδος για τα αυτοκίνητα, γνωρίζαμε την αδυναμία των δοκιμασιών τότε. Αλλά αυτή δεν ήταν μία αδυναμία στον τομέα των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, ε, μάλλον οξυδίου του αζότου, αλλά περισσότερο στον τομέα της κατανάλωσης δοκιμασία κατανάλωση καυσίμου. Ξέρουμε ότι τα αυτοκίνητα χρειαζόταν και κατανάλωναν περισσότερα καύσιμα από ό,τι δείχναν οι επίσημε δοκιμέ. Παρόλα αυτά, η Κομισιόν υποστήριξε τότε την ε, αρμόδια επιτροπή για να δια... δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος δοκιμασιών. Δέκα χρόνια χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτόν τον κύκλο για τα ελαφρά οχήματα αυτό που θα τεθεί το 2017 σε εφαρμογή λοιπόν. Αν το συγκρίνω αυτό με αυτό που έκαναν οι διάδοχοί μου στην Κομισιόν, λέτε ότι χρειάστηκε 10 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς αλήθεια αυτό. Από αυτά τα οποία έχω ακούσει και έχω τα παρτισίδιες πληροφορίες από ό,τι έχετε και εσείς, οι πληροφορίες ξεκίνησαν το 2011. 2011 με 2017 είναι 5 χρόνια. Oh, sorry. Συγγνώμη, λέει Η κυρία Σάλτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όλοι μας νιώθουμε κάποια ματέωση εδώ, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε, να μάθουμε τι έγινε, για να μπορέσουμε φυσικά να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Από τη δική μας πλευρά εσείς ξέρετε ότι υπήρχαν προβλήματα, ανησυχούσατε για τις διατάξεις αναστόλης, αλλά δεν κάνατε τίποτα, γιατί δεν είχατε απόδειξη, είπατε. Εντάξει. Αλλά προσπαθήσατε να φέρετε αυτή τη συζήτηση στην Επιτροπή για την Έγκριση Τύπου, που είναι ένα φόρουμ που περιλαμβάνει και την Κομισιόν και τα μελη Φέρατε τις ανησυχίες σας στην TAAEG, ότι υπήρχε κίνδυνος για χειραγώγηση μέσω διατάξεων αναστολή. Το φέρατε σε αυτή την ε, ομάδα εργασία των εμπειρογνωμόνων. Η απάντηση είναι όχι. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση για το θέμα αυτό, για τις διατάξεις αναστολής στην TAAEG. Γιατί όμως. Ανησυχούσατε. Ξέρατε ότι υπήρχε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά δεν τα φέρατε σε ένα φόρουμ όπου υπήρχε η παρουσία των κρατών μελών και υποτίθεται και η ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Γιατί δεν συζητήθηκε το θέμα αυτό. Δύο εξηγήσει. Πρώτα απ' όλα. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο 2010 για να κατανοήσουμε τι γίνεται. Θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ε, γνώση των πρακτικών έγκρισης τύπου στα διάφορα κράτη-μέλη. Η ομάδα εργασίας αυτή δημιουργήθηκε το 2010 για να έχουμε καλύτερη γνώση για το τι γίνεται από τις ε, ε, επιτροπές έγκρισης τύπου στα κράτη-μέλη οι συζητήσεις στην ομάδα TAAEG γίνονταν πάντα επί τη βάση κάποιου ερωτήματο που τίθετο από τις αρχές έγκριση τύπου ή από τις αρχές του κρατού, των κρατών μελών. Γι' αυτό δεν υπήρξε ποτέ ένα θέμα για αυτές τις... Δεν τέτοιε ποτέ ένα τέτοιο θέμα από καμιά εθνική αρχή ή εποπτική αρχή. Μα μήπως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. εσείς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι. εσείς ξέρατε το πρόβλημα. εσείς ανησυχούσατε, ξέρατε ότι υπήρχε αυτός ο κίνδυνο. Δεν προκάματε. Εντάξει. Πολλοί από εσά έχετε ήδη εμπλακεί στην πρόταση για ένα νέο σύστημα έγκρισης τύπου αλλά εξακολουθείτε να υποστηρίζετε ένα αποκεντρωμένο σύστημα που εναπόκειται στα κράτη-μέλη να κάνουν τα περισσότερα. Αν δείτε το παρελθόν, πιστεύετε πράγματι ότι ένα αποκεντρωμένο σύστημα είναι το βέλτιστο σύστημα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν απάτε στο μέλλον και ότι μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα οχήματα συμμορφώνονται με την ομοθεσία μα. Γιατί εγώ πρέπει να σα πω ότι αμφιβάλλω πολύ γι' αυτό. Αναφέρεστε ίσω στην πρότασή μα, λέει ο κ. Κοζίλο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι υπήρξαν κάποιε βελτιώσει οι οποίε προβλέπονται. Υπάρχουν κάποιες βελτιώσει που προβλέπει η πρότασή μα. Δεν μιλάω για τι ε, διατάξεις αναστολής, γιατί μιλούσαμε για τις, ε, το RDE. Σε ό,τι αφορά αυτή τη μεταρρύθμιση, αν δείτε το κείμενο, βλέπετε ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των ε, εμπλεκομένων είναι πολύ πιο σαφής από ό,τι ήταν στην τρέχουσα νομοθεσία είτε πρόκειται για τις αρχές έγκρισης τύπου, είτε για τις ελληνικές υπηρεσίες, είτε για, τις, για τους κατασκευαστές. Θέλουμε να ενισχύσουμε τα μέτρα εποπτείας της αγοράς με την πρόταση αυτή. Και επίσης θα προβλέπετε για ένα σύστημα αντίδραση των κρατών μελών σε περίπτωση μη συμμόρφωση, κάτι το οποίο δεν προβλέπεται στην τωρινή νομοθεσία. Εισάγει και αποτρεπτικά μέτρα. Εάν οι κατασκευαστές δείξουν ασυνειδησία ή αν οι τεχνικές υπηρεσίες δεν λειτουργούν σωστά και έχει πρόνοιες για κυρώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και υποχρεώνονται οι κατασκευαστές να δίδουν στοιχεία για το λογισμικό των οχημάτων τους και να μπορούν να υπάρχουν εξωτερικοί έλεγχοι. Αυτό προτείνεται. Αυτό το οποίο λέτε είναι γιατί, δεν, γιατί έχουμε ακόμα ένα αποκεντρωμένο σύστημα. Εάν, θα έλεγα εγώ, αν σκεφτούμε τη δυνατότητα να υπάρξει μια ευρωπαϊκή υπηρεσία για αυτά. Αυτό το απορρίψαμε για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί χρειάζεται χρόνο για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κεντρικό φορέας. Και θέλαμε να προχωρήσουμε με ταχύτητα. The cost And the third one... Το δεύτερο είναι το κόστο μιας τέτοια αρχή και τρίτον ότι έχουμε την υποδομή με τις τεχνικές υπηρεσίες και τις αρχές έγκρισης τύπου. Αυτή είναι μια βαριά υποδομή που θα είναι πολύ δύσκολο να αντικαταστήσουμε σε κεντρικό επίπεδο. Θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Αυτή ήταν η λόγια του οποίου δεν ακολουθήσαμε αυτή την οδό. Αλλά λέτε έχουμε ένα σύστημα το οποίο υπάρχει, αλλά δεν λειτουργεί το σύστημα αυτό. Δεν βρήκε τα προβλήματα τα οποία έχουμε ανακαλύψει εδώ. Μήπω είναι καλύτερα να το αναδομήσει κανεί και να φτιάξει ένα νέο σύστημα το οποίο να είναι πιο κεντρικοποιημένο. Εντάξει, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Θα την κάνουμε στην Επιτροπή Εσωτερική Αγορά του Κοινοβουλίου. Συγγνώμη για την ε, παρέμβασή μου. Αλλά το επιχείρημα του χρόνου μέσα σε αυτό το πλαίσιο που το παρουσιάζεται είναι λιγάκι εκτό πραγματικότητα. Κύριε Χένκε. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω ένα ερώτημα προ την κυρία Σιγόφσκα. Είπατε, μάλλον έχετε ακούσει για τις προσπάθειές μας, τις αποτυχημένες προσπάθειες, να προσκαλέσουμε τον τότε Αντιπρόεδρο της Κομισιόν, κύριο Φερχόγεν, στην Επιτροπή αυτή. Και βλέποντας το βιογραφικό σας, βλέπω ότι εσείς έχετε εργαστεί μαζί του, ήσασταν μέρος του γραφείου του, του Γκίντερ Φερχόγεν. Ένα ερώτημα. Θυμόσαστε να έχετε μιλήσει ποτέ στον κύριο Φερχόγεν για τα θέματα που συζητούμε εδώ σήμερα. Η απάντηση είναι σύντομη όχι θυμόσαστε να είχε συζητήσεις με άλλους για αυτό το θέμα, με άλλους φορείς ή επιτρόπους και πάλι πρέπει να πω όχι. Γι' αυτό ίσως πρέπει να τα πω πιο σαφώς. Εργάστηκα με τον Επίτροπο Φερχόγγεν μεταξύ του 2007-2009. Δεν ήμουνα αρμόδια για το χαρτοφυλάκιο αυτό που είναι το αντικείμενο της ακρόασης και ποτέ δεν είχα την ευκαιρία, την ανάγκη ή την ευκαιρία να συζητήσω αυτό το θέμα αυτό ούτε πριν ούτε μετά. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Ζαν, μας στείλατε το βιογραφικό σας. Εκπλήξη μου όμως δεν λέτε τι κάνατε μεταξύ του 2002 και του 2015. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να μας δώσετε αυτές τις πληροφορίες σε μια μεταγενέστερη ευκαιρία, ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει τι κάνατε σε σχέση με αυτά τα οποία συζητούμε εδώ. Ένα θέμα ουσίας τώρα. Όταν η Κομισιόν αποφάσισε τις προδιαγραφές για το Euro 5 και Euro 6, δεν είχατε πληροφορίες όπως πήρατε αργότερα από, τις, ε, από την ομάδα για τα για τις πραγματικές μετρήσεις ελαφρών οχημάτων. Αλλά έχετε τώρα αυτές τις πληροφορίες. Και τώρα, πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί το σύνολο των προδιαγραφών για το Euro 5, Euro 6, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γιατί βλέπουμε ότι το χάσμα μεταξύ των εργαστηριακών ε, μελετών και της πραγματικής, πραγματικών εκπομπών αυξάνεται. Μήπω λοιπόν θα πρέπει να τροποποιηθούν τα πρότυπα για τα ευρώ 5 και ευρώ 6. Αν το ερώτημα είναι αν εργαζόμαστε τώρα σε νομοθεσία για, για μια κατηγορία ευρώ 7 οχημάτων, η απάντηση είναι όχι. Αυτό το οποίο όμως προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι ο ενοποιημένος κύκλος ελέγχου, το WLTP, η RDA και επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των οχημάτων. Λοιπόν, τα περισσότερα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους μας έχουν μια ηλικία περίπου 2 ετών, μερικών ετών, 7-8 χρόνια είναι η μέση ηλικία τους ίσως. Τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι μια δοκιμασία η οποία δείχνει καλά αποτελέσματα όταν το αυτοκίνητο είναι καινούριο και βγαίνει για πρώτη φορά στον δρόμο, εξακολουθούν όλα αυτά να ισχύουν μετά από κάποια χρόνια χρήσης, πραγματικής χρήση στον δρόμο. Η απάντηση σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι ένα ουσιώδες ερώτημα. Όπως ξέρετε πολύ καλά, η νομοθεσία σήμερα βασίζεται στην ε, ε, εξέταση των οχημάτων όταν τίθενται σε κυκλοφορία, αλλά είναι κάπως αδύναμη για να ελέγξει την κατάσταση των αυτοκινήτων όταν είναι σε κυκλοφορία για κάποιο διάστημα. Το πακέτο αυτό το οποίο συζητούμε σήμερα για την έγκριση τύπου και την νομοθεσία RDE δίνει ακριβώς την απάντηση στο ερώτημα σας αυτό λέγοντας ότι θα δημιουργήσουμε ε, δοκιμασίες ελέγχου των οχημάτων εν κυκλοφορία από την ε, Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και αυτό θα γίνει και με την αρρωγή του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Όπω είναι και με την έγκριση τύπου και έχουμε σαν πρόθεση να αναπτύξουμε περισσότερο αυτή την έννοια για το τρίτο πακέτο, οπότε θα κάνουμε ελέγχου εν κυκλοφορία των οχημάτων για τη συμμόρφωσή τους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι εν επεξεργασία. Φέντελε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ακρόαση και Έχω ζητήσει ορισμένε πληροφορίε πολλέ φορέ στι ακροάσει. Έχουμε μιλήσει για την ημερομηνία που ξεκίνησαν αυτέ οι διαδικασίε στην Κομισιόν και για το γιατί έχουν καθυστερήσει. Θυμάμαι συζητήσει με την ε, Υπηρεσία Περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είπαν ήδη το 2004 σε μια έκθεσή του ότι υπήρχαν τεράστιε αποκλήσει μεταξύ των εκπομπών όπως υπολογιζόταν και των πραγματικών εκπομπών. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε πίσω το 2004. Έχουμε μια έκθεση η οποία υποδεικνύει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τις εκπομπές. Βρισκόμαστε τώρα στο 2016, έχουν περάσει 12 χρόνια και παρόλα αυτά ακόμα δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την νομοθεσία η οποία έχει θεσπιστεί. Μετά από αυτά που είπε και ο συνάδελφός μου από τους σοσιαλιστές προσπαθώ να φτάσω στην ουσία του θέματος. Τι πήγε στραβά, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί το πρόβλημα αυτό και γι' αυτό θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα, όχι για τι διαδικασίε, αλλά για την ε, ισορροπία των δυνάμεων και την νομοθεσία. Θα λέγατε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με την ε, κατανομή εξουσιών μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιών για αυτή την νομοθεσία. Είναι δύσκολο για μένα να εκφέρω προσωπική γνώμη εδώ. Αλλά νομίζω το ζήτημα δεν είναι τόσο η ισορροπία των αρμοδιοτήτων ή της εξουσίας ανάμεσα, της, ε, ανάμεσα στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ωστόσο, το σύστημα που έχουμε σήμερα για την συγκρίση τύπου και τη σχετική νομοθεσία δεν είναι ικανοποιητικό, είναι υπερβολικά επίκες και αυτό είναι ένας από τους λόγους που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει την τροποποίηση του. Οι προτάσεις μας για τη μεταρρύθμιση του εστιάζονται σε ακριβώς εκείνα τα σημεία που θέλουμε να βελτιώσουμε. Για παράδειγμα, η αποπτία των κατασκευαστών να μην γίνεται μόνο από ένα κράτος μέλος, αλλά να αυξηθεί και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην όλη διαδικασία, καθώς επίσης να προβλέπεται ότι οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όχι μόνο στο εθνικό, ότι θα υπάρχουν πιο συχνά αναφορέ όσον αφορά την υλοποίηση τη νομοθεσία από την πλευρά των κρατών μελών. Αυτά είναι τα ζητήματα που κατά την άποψή μου πρέπει να βελτιωθούν και τα σημαντικά, όχι τόσο ισορροπία μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Γνωρίζατε την έκθεση της EEA από το 2004 που αναδείκνυε τα προβλήματα. Um, sorry, it's a long time ago and I'm... Um, Αυτό έχει συμβεί πριν πολύ καιρό και δεν μπορώ να θυμηθώ εάν το 2004 είχα διαβάσει μια έκθεση. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι είχαμε υποβάλει προτάσεις για τη μείωση των εκπομπών οξυδίου του αζότου και αν θα θυμάστε η Επιτροπή είχε αρχικά προτείνει μόνο το Euro 5 και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επέμειναν να υπάρξει και μια πιο αυστηρή νομοθεσία, ε, το Euro 6 κάτι το οποίο υποστηρίξαμε και εμείς και τελικά εγκρίθηκε. Όμως θέλω να είναι ξεκάθαρο ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης, το οποίο είναι ότι οι εκπομπές οξυδίων του αζότου είναι υψηλότερες από όσες θα θέλαμε, από θα έπρεπε. Αυτό συζητούσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν συζητούσαμε τις διατάξεις αναστολής. Ερώτηση γίνεται όλο και πιο σαφές σε εμένα ότι το σύστημα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι υπερβολικά περίπλοκο και δεν ε, έχει τους κατάλληλους μηχανισμούς. Υπήρχε ε, η έκθεση του 2014 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που αναδείκνυε τα προβλήματα και δεν ε, ελήφθησαν μέτρα για την αντιμετώπιση τους. Επομένως εδώ έχει συμβεί ένα σφάλμα, ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να διορθώσουμε. Και το ερώτημα μου είναι Ποιε διαδικασίε θα έπρεπε να ακολουθούνται όταν υπάρχει μία έκθεση η οποία λέει ότι η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται. Για οποιονδήποτε λόγο, είτε είναι για τις ε, διατάξεις αναστολής, είτε εξαιτία των ορίων που τίθενται. Για να λειτουργεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία, για να υπάρχει ευρωπαϊκή συνεργασία, πρέπει να εξασφαλίζουμε την υλοποίησή της. Είχαμε εδώ λοιπόν μια έκθεση ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. Και το ερώτημά μου είναι ποιο μηχανισμό, ποια διαδικασία πρέπει να εγκαθιδρύσουμε έτσι ώστε να εξασφαλίζουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας που εγκρίνουμε ως συνομοθέτες. Η Επιτροπή. Θα μιλήσω ως άνθρωπος που είναι ε, με το ένα πόδι έξω από αυτήν την διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση και αυτή η οργή στην ε, εξεταστική σας επιτροπή. Όσον... Γιατί υπάρχει αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διερεύνησε τη χρήση των διατάξεων αναστολής. Αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος, Το γνωρίζω, θα έπρεπε, θα θέλατε να ε, έχει δραστηριοποιηθεί περισσότερο ή πιο γρήγορα η Επιτροπή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που συζητούμε είναι τι έκανε η Επιτροπή και τι θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος. Και σε αυτό το θέμα, στο δεύτερο, ως εξωτερικός παρατηρητής, τρέψτε μου να πω, ότι εξεπλάγει θετικά, εντυπωσιάστηκα, με το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να υποβάλει μια πρόταση λίγες ημέρε μετά τη δημοσιοποίηση του σκανδάλου της Volkswagen. γνωρίζουμε ότι η νομοθεσία σχετική είχε, ε, το πρώτο μέρος της είχε ήδη εγκριθεί πριν την δημοσιοποίηση του σκανδάλου της Volkswagen. Επομένω πιστεύω ότι είναι άδικο να λέμε ότι η Επιτροπή αδράνησε. Πιστεύω ότι ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιήθηκε η Επιτροπή είναι ακριβώς ο σημαντικότερος, είναι εκείνο που θα εξασφαλίσει ότι τέτοια προβλήματα δεν θα υπάρξουν στο μέλλον. Και η νομοθεσία με την, ε, ε, την οποία ε, εγκρίνεται πρέπει να καλύπτει χιλιάδες διαφορετικές υποθέσεις και περιπτώσεις. Ε, να μην ε, περιοριστούμε, να μην εστιαστούμε μόνο σε αυτό το μεμονωμένο περιστατικό που ήταν η χρήση μιας συγκεκριμένης διάταξης αναστολής που αποκαλύφθηκε το 2015. Έχουμε την εξή ερώτηση να θέσω. Αυτή τη, φορά, αυτή τη στιγμή ακούμε από τέσσερις υπαλλήλους της Επιτροπής να μας λένε όμορφες ιστορίες, ενώ ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως θεσμικό όργανο έχει αρνηθεί να μας παράσχει τα ε, έγγραφα που έχουμε ζητήσει. Ζητήσαμε έγγραφα από το 2011 ως το 2013 και λάβαμε 7 σελίδες. Πλάκα μας κάνετε. Υποτιμάτε την νοημοσύνη μας. Το είναι σίγουρο ότι έχετε ανταλλάξει εκατοντάδες email και επιστολές την περίοδο 2011-2013 που ήταν ακριβώς η περίοδος που η αυτοκινητοβιομηχανία προσπαθούσε να μην υιοθετηθεί το PEMS. Επομένως δεν μπορώ να δεχτώ να έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αρνείται να μας παρασχεί έγγραφα έτσι ώστε να, μπορούμε να, μην, να μπορούμε να ελέγξουμε την αλήθεια αυτών που μας λένε οι υπάλληλοι της. Επίσης, κύριε Ζαν, μας είπατε ότι τον Ιούνιο του 2014 θα έπρεπε να ληφθεί η απόφαση για τους συντελεστές συμμόρφωσης. Και δεν προχώρησε αυτή. Η συζήτηση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014, δεν προχωρούσε και 10 μέρε μετά την δημοσιοποίηση του σκανδάλου του Volkswagen καταλήξαμε σε απόφαση. Πράγμα που αποδεικνύει ότι ήταν το σκάνδαλο του Volkswagen που μα κινητοποίησε τελικά. Επανέρχομαι λοιπόν σε μια, ε, ένα email, με το, μάλλον επιστολή του 2008, με την οποία ζητείτε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών να μετρήσει η Γενική Διεύθυνση επιχειρηματικότητα τους διζηλοκινητήρες που εξάγονται στις ΗΠΑ. Και το ερώτημά μου είναι το εξή. Η Γενική Διευθύνση Περιβάλλοντο το ζήτησε αυτό από το JRC, από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το 2008. Είχε την περιέργεια τότε λοιπόν, το 2008, ε, να μάθει η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ποια τεχνολογία θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να τηρηθούν τα αυστηρότερα ε, όρια των Ηνωμένων Πολιτικών. Το οποίο μας δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, γνωρίζει κάτι και το ζητάει αυτό το JRC. Και το ερώτημά μου είναι, έγινε αυτή η μελέτη. Εάν πότε και αν όχι γιατί. I Οι συνάδελφοι που παρευρίσκονται εδώ είναι από την Γενική Διεύθυνση ανάπτυξη, τη UGROW και δεν μπορούμε να απαντήσουμε εκ μέρου τη γενική Διεύθυνση περιβάλλοντο. Νομίζω ότι την απάντησή σα καλύτερα θα τη λάβετε από αυτό εκείνον που έστειλε ή εκείνον που έλαβε αυτή το, αυτό το μήνυμα. Όλοι γνωρίζουν ότι η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος είχε δικαίωμα να ζητήσει από το JRC να, να κάνει μια μελέτη. Αλλά το JRC εξαρτάται από εσά. Είμαι σίγουρος ότι όταν λάβουμε τα email που έχουμε ζητήσει επιτέλους στην κατοχή μας, θα αποδειχθεί ότι ψεύδεστε. Γιατί θα με εξέπλητε η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος να μην έχει κοινοποιήσει το αίτημά της και σε εσάς. όταν γνωρίζουν ότι έτσι και αλλιώς εσείς πρέπει να εγκρίνετε την διενέργεια της μελέτης από το JSC, από το Κοινοκέντρο Ερευνών. Απάντηση της Επιτροπής. Εγώ δεν ενθυμούμαι αυτή την ανταλλαγή μηνυμάτων. Μπορώ να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ε, το διερευνήσω και να ε, σας δώσω τα σχετικά στοιχεία στην Επιτροπή σας. Ωραία, ας επιστρέψουμε το 2007-2008. Πότε ακριβώς διενήργησε τους ελέγχους για τα ε, οχήματα Euro 5 το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Πότε ακριβώς, γιατί μετρήθηκαν οι εκπομπές ε, σε αυτά τα 14 οχήματα. Πότε ακριβώς μέσα στο 2009. Αρχές, μέσα, τέλος. And Και μου μην πείτε ότι δεν θυμάστε, γιατί τότε ήταν ε, σκάνδαλο όλο αυτό. Ε, είχε τεράστια, ε, τεράστια πίστη στην κοινή Δεν θυμάστε πότε έγιναν αυτά, αυτά τα τεστ. Μα τι είναι αυτά τώρα. Η Κομισιόν. Τα τεστ αυτά έγιναν την περίοδο 9-10, για τα οποία λάβαμε έκθεση από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Πότε ακριβώς, είναι η ερώτηση. διότι έχω την εξή εντύπωση. Τα τεστ στο Κοινό Κέντρο Έρευνας έγιναν, εκπονήθηκε η μελέτη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνιστικότητας απαγόρευσε τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτών των τεστ. Και αυτό πρέπει να είναι τέλη του 2009, αρχές του 2010. Χάσαμε πάνω από ένα χρόνο μετά την ε, διεξαγωγή των τεστ. Με δική σας ευθύνη. Πρόεδρος, αν δεν θυμούνται ε, μπορούν να μας δώσουν γραπτή απάντηση. Μα δεν μας στέλνουν τα email από εκείνη την περίοδο λέει ο κύριος βουλευτής. Πρόεδρος. Α, όχι, εκπρόσωπος Κομισιόν. Δεν μπορώ να σας πω τον ακριβή μήνα πότε ξεκίνησαν τα τεστ από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η μελέτη του 2010, το πρώτο τμήμα που δημοσιεύθηκε το 2011, το πρώτο τμήμα έγινε μετά από συγκεκριμένο αίτημα των συναδέλφων στη Γενική Διεύθυνση επιχειρηματικότητα το αίτημα να γίνουν αυτά τα τεστ και να γίνει η μελέτη ήταν από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας Enterprise το 9. Το κοινό κέντρο ερευνών έλεγξε σε δύο ομάδες τα οχήματα. Η πρώτη, η, η πρώτη φουρνιά ήταν 11 και η δεύτερη άλλα 3 αλλά προσπαθούσαν να εξετάσουν διαφορετικά οχήματα, όχι μόνο diesel, αλλά και βενζινοκίνητα και υβριδικά. Και η μελέτη δημοσιεύθηκε κατόπιν. Δημοσιεύονταν σταδιακά μόλις ε, προέκυπταν. Όπως σας είπα, τα τεστ έγιναν 2009 και η έκθεση δημοσιεύθηκε το 2011. Εσείς ε, εμποδίσατε την νωρίτερη δημοσίευση των μελετών. Υποχρεώσατε να διοργανωθεί ένα workshop από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και επειδή φοβόσταν τόσο πολύ τα αποτελέσματα των τεστ, αποφασίσατε να επινοήσετε αυτή, τη μελέτη, αυτή την ομάδα εργασίας RDE για να δείξετε ότι δίθεν έχετε κάνει κάτι όταν θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Πρόεδρος, απαντήστε ναι ή όχι. Οπωσδήποτε όχι, λέει η Κομισιόν. Σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Τη συζήτηση για την πρόσβαση στα έγγραφα την έχουμε ήδη κάνει. Θα την ξανακάνουμε το απόγευμα, όπου οι συντονιστέ θα συζητήσουν τα θέματα εμπιστευτικότητα. Αλλά θα ασκήσουμε πολύ έντονη πίεση σε πολύ υψηλό επίπεδο, κύριε Τούρμες, για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα πρόσβασης στην ε, τεκμηρίωση. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, όχι άλλο. Ο κύριος Τζούλο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, μιλήσαμε για ε, την εντιμότητα που πρέπει να υπάρχει διαδικασία. Θέλω να θέσω την εξή ερώτηση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε τόσο καιρό για να υπάρξει ο καθορισμός αυτής της νέας διαδικασίας. Σε μία πρόσφατη μελέτη αποδεικνύεται ότι οι μετρήσεις διοξιδίου του άνθρακα με αυτό το σύστημα θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ε, ελλειπείς, θα υποτιμούν ε, τις διαστάσεις του προβλήματος. Γιατί να μην ε, επιλέξουμε τον κύκλο οδήγησης τεμής για να έχουμε καλύτερη εκτίμηση, όπως ακριβώς είχε προτείνει και ο Ευρωπαϊκός Φορέας Περιβάλλοντος. Και η διαδικασία αυτή, όπως ξέρετε, έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα σχόλιο πριν απαντήσω στην ερώτησή σα. Κοιτάξτε. Για τα έγγραφα. Σας έχουμε αποστείλει μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 129 έγγραφα. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα εμπιστευτικότητα, αλλά δεν ισχύει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εντύπωση ότι σας στείλαμε μόνο 7 έγγραφα. Στείλαμε σχεδόν 130. Σας παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος, δεν θα κάνουμε τώρα διάλογο. Σας παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Τώρα για τον WLTP δεν μπορώ να απαντήσω. WLTP θα σας δώσουμε γραπτή απάντηση. Γιατί κανείς από εμά ε, δεν έχει αυτή τη στιγμή ε, τα στοιχεία. Ωραία, θα πάρουμε γραπτή απάντηση, λέει. Παρακαλώ, συνεχίστε. Α, εντάξει, τελειώσατε. Ωραία, ωραία. Ωραία, λίγη ο δεύτερος γύρος. Τώρα τελευταίος γύρος ομιλητών. Τρία λεπτά παρακαλώ. Έχουμε κάποια καθυστέρηση. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να τηρείτε το χρόνο σας. Ο κύριος Νίντεμάια. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Δύο ερωτήσει. Πρώτη. Ε, είναι βέβαια τώρα και μια άλλη προκατακτική ερώτηση. Είστε κι εσείς τόσο απογοητευμένοι όπως και εμείς, αλλά δεν περιμένω απάντηση. Τώρα, αναφερθήκατε σε προηγούμενες μετρήσεις ε, μέτρηση της κατανάλωσης και του δεξιδίου του άνθρακα και ξέρουμε ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές για αυτές τις δύο παραμέτρους μεταξύ εργαστηριακών και πραγματικών συνθήκων ορισμένες έχουν να κάνουν με τον τρόπο οδήγηση, άλλοι έχουν να κάνουν με αντικειμενικού παράγοντε, αλλά ξέρουμε εδώ και χρόνια τι προσαρμογές κάνουν οι κατασκευαστές. Για παράδειγμα υπάρχει μία έκθεση που λέει προσέξτε την διαφορά επίπεδου με το 2003, από το 2003 και επίσης και ένα ε, άρθρο είδα στο BBC για το τι προσαρμογές κάνουν οι κατασκευαστές όταν ελέγχονται τα οχήματά τους. Άρα δεν μπορούμε να πούμε πως δεν υπήρχαν στοιχεία. Και ως επίπτωση ακριβώς ε, αυτών των προσαρμογών τα αποτελέσματα ήταν παραπλανητικά. Πείτε μου παρακαλώ τι κάνατε τότε, πώς αντιδράσατε ω Κομισιόν και τι θα κάνουμε για να μην επαναληφθεί αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Και δεύτερον, για αυτού τους μηχανισμούς αλλίωσης. Υπάρχουν πολλά είδη τέτοιων μηχανισμών και αν δείτε τι έχει γραφτεί τα τελευταία χρόνια θα δείτε ότι υπήρχαν σοβαρέ υποψίε για πολύ πιο απλοϊκούς ε, μηχανισμούς από αυτούς που χρησιμοποίησε η Volkswagen. Για παράδειγμα, έλεγχαν τη θερμοκρασία, το αν κουνιόταν το τιμόνι, αν ε, είχε ε, ε, ε, σβήσει το GPS. Και όλα αυτά ήταν η λεγόμενη στρατηγική εκπομπών του κινητήρα. Τα εξετάσατε όλα αυτά στο παρελθόν. Αν υπήρχαν στοιχεία ότι προσπαθούσαν οι κατασκευαστές να είναι διαφορετικές οι εκπομπές στα εργαστηριακά τεστ από τις πραγματικές συνθήκες. Ευχαριστώ πολύ. Για το πρώτο σας ερώτημα, <clears throat> διαφορές μεταξύ κατανάλωσης ε, καυσίμου και εκπομπών διοξιδίου Τι έχουμε κάνει για αυτά. Εμείς βασιστήκαμε στο έργο που έχει γίνει στο φόρουμ των, του ΟΗΕ στη Γενέβη, που ξεκίνησε το 2009 στην πραγματικότητα. Το 2014 εγκρίθηκε η κατάλληλη νομοθεσία, οπότε έχουμε τον κανονισμό που προβλέπει νέους ε, τρόπους δοκιμασίας που είναι πιο επακριβείς για τις εκπομπές διοξιδίου του Άνθρακο. Αυτός ο μηχανισμός έχει περάσει σε νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα σε δύο χρόνια. Την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσε αυτή η διαδικασία και θα αποσταλεί στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για έλεγχο είναι σαφέ λοιπόν, ξέραμε ότι υπήρχαν διαφορέ, αμέσω λάβαμε δράση και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε μεταγράψει αυτό στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τελειώσει εδώ αυτή η διαδικασία, θα τεθεί σε εφαρμογή και εμεί θα παρακολουθήσουμε τι μετρήσει διοξιδίου του άνθρακο. αν υπάρξουν ανάγκε να προχωρήσουμε περισσότερο, γιατί και ο έλεγχος, ε, το σύστημα WLT είναι και αυτό έλεγχο <clears throat> εργαστηρίου, θα προχωρήσουμε. απλώ το ερώτημά μου. Αυτό σημαίνει ότι οι μετρήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν ήτανε, ε, έχουν διακριβωθεί παρανομίες ή όχι. Όχι, δεν θα ήταν παράνομες αυτές οι μετρήσεις που έγιναν στο παρελθόν. Οι τωρινές συνθήκες, ε, ε τα τωρινά όρια βασίζονται στις συνθήκες μέτρησης που ακόμα εξακολουθούν να είναι ε, έγκυρες. Τώρα προσπαθούμε να βρούμε τις νέες διαδικασίες ε, για την ε, μέτρηση, θα παρουσιαστούν προτάσεις αυτές για τη μεταβατική περίοδο θα υπάρξει ένα είδος ισχυωτισμού μεταξύ των δύο συστημάτων. Από το 2018 θα πρέπει να γίνεται η έγκριση τύπου με τη νέα διαδικασία. Ναι. Ο κύριος Ζουρίνιου. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μια έκθεση αντικτύπου για το RDE ήδη από το 2013. Εσείς επιμένετε ότι δεν είχατε κανένα στοιχείο ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής για χειραγώγηση των εκπομπών, αλλά υπάρχει μια μελέτη που αξίζει τον κόπο να σας υπενθυμίσω. Θα το διαβάσω στα αγγλικά γιατί δεν έχω το κείμενο στα γαλλικά. αυτής της μελέτης. Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις για παράνομες πρακτικές από διάφορους ε, κατασκευαστές για τη χρήση των συστημάτων ε, κατά της ε, ρήπανσης για να βελτιώσουν την απόδοση των οχημάτων. Και εσείς λέτε ενώπιον αυτού ότι δεν υπήρχαν καθόλου στοιχεία. Είναι σαν να λέτε ότι αυτή η μελέτη δεν είναι αξιόπιστη για σας. Δεν είναι αξιόπιστη αυτή η μελέτη. Τότε γιατί χρησιμοποιήθηκε από την Κομισιόν για να αναφέρει στα κρατημέλη ότι υπήρξαν παραδιάσει σε σχέση με τα όρια των εκπομπών οξυδίου του αζότου. Γιατί υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτή η μελέτη δεν οδηγεί σε συνέπειες για την Κομισιόν, αλλά έχει συνέπειες ό,τι αφορά τον έλεγχο των κρατών μελών. Αυτό το οποίο ήταν το πιο σημαντικό για μας ήταν η αποφασιστικότητα που είχαμε να αλλάξουμε τη μέθοδο ελέγχου των εκπομπών. Η διαδικασία η οποία ήταν εν εφαρμογή τότε και εφαρμόζεται ακόμα για μας δεν έπρεπε να τροποποιηθεί παρά μόνο με ριζικό τρόπο χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική άποψη. Η έκθεση που αναφέρεται ήταν ένα πρόσθετο στοιχείο το οποίο καταδεικνύει ότι ήταν πραγματικά κατεπήγον να αλλάξουμε τη διαδικασία ε, μέτρηση των πραγματικών εκπομπών. Ναι. Αλλά εσείς ξέρατε ότι υπήρχαν ε, διατάξεις αναστολής ή όχι. Εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν το ξέρατε τότε. είχαμε τη γνώση του γεγονότος ότι ήταν απαγορευμένες, αλλά και ότι δυνητικά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό το νέο σύστημα RDE έχει σαν στόχο να μειώσει συστηματικά την δυνατότητα χρήσης αυτών των απαγορευμένων καρπών. Κύριε Ζωρίνιο, εκτός μικροφώνου. Μικρόφωνο παρακαλώ μπορώ να συμπεράνω ότι εσείς ξέρατε ότι υπήρχαν διατάξεις αναστολής που χειραγωγούσαν τις εκπομπές και αυτό είναι το όνομα. Με κάποιο τρόπο, με κάποιο όνομα το ξέρατε ότι υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Ο κίνδυνος υπήρχε. Και ξέραμε ότι υπήρχε ο κίνδυνος, λέει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Κύριε Γκαλπέλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. εμείς νιώθουμε μία ματέωση. Θα θέλαμε να έχουμε πληροφορίες αξιόπιστες πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να βασιστούμε. Δεν είναι η δική μας Επιτροπή η οποία έχει ζητήσει πληροφορίες ε, αλλά είναι υποχρέωση Κομισιόν <clears throat> να παράσει αυτές τις ε, πληροφορίες. Οι πληροφορίες οι οποίες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες δεν καθιστούν δυνατό, δείχνουν ότι δεν ήταν δυνατόν να αποφευθεί αυτό το σκάνδαλο. Τελικά χρειάζεται να υπάρξει ένα σκάνδαλο για να μπορέσει η Κομισιόν να κινητοποιηθεί και να τροποποιήσει την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω μια πολύ ε, δυσάρεστη αίσθηση από αυτά τα οποία έχετε αναφέρει. Το ερώτημα μου τώρα το εξής. Η ομάδα πυρογνωμόνων που είναι αρμόδια για την έγκριση τύπου τι θα μπορούσε να επιτύχει η, τι μπόρεσε να επιτύχει αυτή η ομάδα σε στο επίπεδο της εναρμόνισης των ε, εγκρίσεων τύπου στα κράτη-μέλη. Ο κανονισμός 715 του 2007 τώρα, σε ό,τι αφορά τις ε, ε διατάξεις ε, αναστολής. Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία περιλαμβάνε και σε ποιο βαθμό μπορούσαν οι κατασκευαστές να τα ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο. Αναφερθήκατε ότι και αυτός είναι ένας κανονισμός ο οποίος πρέπει να τροποποιηθεί. Έχετε κάνει όμως τις απαραίτητες ενέργειες για να ξεκινήσει η αλλαγή αυτού του κανονισμού. Και το τελευταίο μου ερώτημα έχει και πάλι να κάνει με τις ε, διατάξεις αναστολής. Ο ορισμός που δίνεται για αυτές τις συσκευές στις ΗΠΑ είναι πολύ διαφορετικός από αυτός που αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διάφορε διάφορες ΜΚΟ έχουν ε, επιβεβαιώσει ότι ε, πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Μπορείτε να αναφερθείτε στα πλέον και τα μειονεκτήματα τουρισμού σας. Ευχαριστώ. Για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση πρέπει να σας πω πρώτα ότι εμείς θέλουμε να εισαγάγουμε αυτό, αυτή τη δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες που μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο διατάξεων αναστολής. Το δεύτερο σημείο το οποίο αναφέρθηκε και πρέπει να υπογραμμαστεί είναι ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να δημοσιοποιούν την στρατηγική ελέγχου των εκπομπών που ακολουθούν και θα υπάρχει και αυτό είναι στην ε, μεταρρύθμιση της διαδικασίας έγκρισης τύπου, θα πρέπει να υποβάλουν το λογισμικό τους στις αρχές έγκρισης τύπου, ώστε να είναι δυνατόν να γίνονται ανεξάρτητοι έλεγχοι και έλεγχοι σε οχήματα εν κυκλοφορία. Το άλλο θέμα, η συνάδελφος, είπατε ότι δεν είναι σαφής η ορισμοί στον κανονισμό 715-2017. Είναι πολύ σαφής ο κανονισμός και μπορεί να εφαρμοστεί ήδη και, και τώρα από τις αρχές και τους κατασκευαστές. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια κοινή ερμηνεία και σε σχέση με τους κανόνες των Ηνωμένων Πολιτειών, η νομοθεσία των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ παρόμοιες. Βασίστηκε στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Η διαφορά είναι στη συνέχεια που δίνεται. Με την δήλωση, παραδείγματος για τη στρατηγική που ακολουθούν οι κατασκευαστές του κινητήρα και επίσης χρειάζεται μια διευκρίνηση για το πώς να εφαρμόσει την νομοθεσία. Κατά άλλα είναι η ίδιοι νόμοι. Oui, je voulais savoir... Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή για την ομάδα εμπειρογνωμόνων και τον εσωτερικό της κανονισμό. Προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό της TAAEG να υποβάλει η Κομισιόν προτάσεις. Η απάντηση είναι ναι. Ωραία. Τότε, σκεφτήκατε ποτέ την πιθανότητα ή μήπως το κάνατε κιόλα να ζητήσετε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη μια συζήτηση για την εφαρμογή των άρθρων 5 και 13 του κανονισμού 715, έτσι ώστε να συζητηθεί το θέμα με τους εκπροσώπους των κρατών μελών, να μάθετε τι είχαν πράξει και τι όχι, και πιο συγκεκριμένα, τι συνέχεια δώσατε στην επιστολή της Κομισιόν που αναφέρεται στην νεκροπτή ερώτηση 8 όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων 5 και 13. Απάντηση της Επιτροπής. Πράγματι είχαμε προβλέψει στην ημερησία διάταξη συζητήσεις ε, για την κανονισμό 715 και για τις διατάξεις αναστολής υπό την ευρεία έννοια αν θέλετε. Έγινε μια συζητήση τον Οκτώβριο πέρυσι, το Φεβρουάριο και άλλη μια την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα όπου συζητήσαμε τα θέματα που σχετίζονται με αυτές τις με τις πρακτικές, τον ορισμό, να καταλήξουμε σε μια κοινή ερμηνεία του ορισμού. Δηλαδή ζητήματα που ακριβώς αυτό το φόρουμ έχει την αρμοδιότητα να συζητά. Ερώτηση. Όμως η επιστολή της Επιτροπής προς είναι πολύ παλαιότερη από τις συναντήσεις που μας αναφέρατε και θα ήθελα να γνωρίζω αν είχε συζητηθεί το θέμα στην TAAG, στην ομάδα εμπειρογνωμόνων, πιο νωρί. Απάντηση. Όχι, δεν έγιναν τέτοιες συζητήσεις για την ερμηνεία του κανονισμού γύρω 5, γύρω 6 κατά την ε, περίοδο 2012, 2013 και 2014. Μάλιστα, δηλαδή πρόκειται για έναν κανονισμό του 2007 και περιμένετε το σκάνδαλο του Volkswagen για να το θέσετε το ζήτημα στην ημερήσια διάταξη και να το συζητήσετε ακριβώς στο φόρουμ το οποίο προβλέπετε ε, για την ανταλλαγή απόψεων με τις ε, αρχές των κρατών μελών και δεν το κάνατε πιο νωρίς. Αυτό μας λέτε. Οι συζητήσει για τα διατάξει αναστολής έγιναν στην TCMV κατά τη διάρκεια του 2014. Στο πλαίσιο ακριβώ θα συζητήσουμε για την υλοποίηση του κανονισμού γυρω 5 6. Ερώτηση. Ναι, αλλά εγώ εστιάζω στα άρθρα 5 και 13 του κανονισμού 7 7-15. Ε, αυτό ήταν το αντικείμενο της ερώτησης μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. και εμένα το ερώτημα μου έχει σχέση με τον κανονισμό 715 του 2007. Στο άρθρο 5 δάφιο 2 αναφέρονται ε, εξαιρέσεις, περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση αυτών των διατάξεων αναστολής. Αναστολής του συστήματος ε, ελέγχου εκπομπής καυσαερίων και η πρώτη περίπτωση που αναφέρεται είναι η προστασία του κινητήρα όταν αυτή είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του αυτοκίνητου. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι ακριβώς ε, καλύπτεται εδώ, συγκεκριμένες περιπτώσεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι έτσι όπως διατυπώνεται το άρθρο είναι υπερβολικά ευρύ. Τι ακριβώς ε, επιδιώκουμε εδώ, πώς θα έπρεπε να το ερμηνεύσω αυτό το σημείο του κανονισμού. Παναλαμβάνω, άρθρο 5, παράγραφος 2, ε, υποσημείο α. Η Επιτροπή σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα τέτοιων εξαιρέσεων. Και θα μπορούσαμε να σας δώσουμε και περισσότερα στοιχεία για το πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια εξαίρεση. Το προφανές που μου έρχεται στο μυαλό είναι όταν γίνεται προσπέραση. Τότε χρειάζεται πλήρη, η πλήρης ισχύ του κινητήρα. Και σε αυτήν την περίπτωση επιτρέπεται να ε, απενεργοποιηθεί προσωρινώς το σύστημα ελέγχου εκπομπής καυσαέριων. Αυτό είναι μία από τις πιθανές εξαιρέσεις, οι οποία βέβαια πρέπει να εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και πολύ περιοριστικά δηλαδή. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που είχα, Μπορώ να σας δώσουμε, μπορούμε να σας στείλουμε γραπτά και άλλα. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση για τον κύριο Σούλτε Μπράουκ, ο οποίος από ό,τι ακούσαμε είναι ήδη συνταξιούχος. Ωραία, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Όταν ε, το 2007 εγκρίναμε τους τύπους 5 και 6, ε, υποχρεωθήκατε να δείτε και τα τεστ. Και η ομάδα εργασία το 2011 ξεκίνησε να λειτουργεί. Γιατί ενώ από το 7 πρέπει να ελέγξετε, μόνο το 11 άρχισε να λειτουργεί αυτή η ομάδα. Ο κύριος Φίλιπ Ζων ήταν υπεύθυνο γι' αυτό επειδή εγώ είχα αναλάβει άλλα καθήκοντα και έχει απαντήσει. Ο κανονισμός λέει συγκεκριμένα ότι η νέα διαδικασία ελέγχου για τα 5 και 6, γύρω 5 και 6, θα πρέπει να καθορίσει οριακές τιμές. Δηλαδή έπρεπε να έχουμε τα οχήματα να κυκλοφορούν, τα οποία θα έπρεπε να τηρούν αυτά τα όρια. Και τα οχήματα αυτά άρχισαν να κυκλοφορούν από το 9-10. Μα τότε ήδη το 2009 θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει να λειτουργεί αυτή η ομάδα εργασία. Ναι, αλλά εξηγήσαμε ότι ήδη το κοινό κέντρο ελέγχου ξεκίνησε τα τεστ το 2009 και μόλις είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτών των τεστ από ό,τι καταλαβαίνω συστήθηκε αυτή η ομάδα εργασίας. Η Επιτροπή μας έχει την εντύπωση παρόλα αυτά ότι δεν εργαστήκατε με την αναγκαία ταχύτητα. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος γιατί ο, για τον οποίο ο Επίτροπος Φερχόγγεν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για αυτά τα θέματα, αρνήθηκε να παρευρεθεί. Γιατί βέβαια ο κύριος Φερχόγγεν θα ήταν ο αρμόδιος για να απαντήσει και παρόλα αυτά δεν ήρθε. μήπως θα μπορούσαμε να καλέσουμε την επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του ή κάποιους άλλους. Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έρθει εδώ ο ίδιος ο Επίτροπος κ. Φερχόγκερ. Νομίζω ότι τα ερωτήματα που θέτετε τα έχει απαντήσει αναλυτικά ο συναδελφός μου Φιλίπ Ζων ήδη. Σας ρώτησα εάν υπάρχουν άλλοι οι οποίοι αν δεν θέλουν τώρα όπως για παράδειγμα ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικότητας, είτε διευθυντές, είτε τμήματάρχες. Ε, μήπως θα μπορούσατε να μου προτείνετε τα ονόματα, δεν θα τα πείτε, δεν θα μου τα γράψετε τώρα απ' έξω. Ίσως ο συνάδελφός σας Φιλίπ Ζων θα μπορούσε να μας προτείνει. Όχι, λέει ο κύριος Φιλίπ Ζων, δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να σας δώσουμε τέτοιες πληροφορίες. Και επίσης υπάρχει και ένα θέμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Ντάντε. Ντάντι. Ευχαριστώ. Εγώ πραγματικά παραμένω έκπληκτος από ότι το 1 τρίτο των ελέγχων συμμόρφωσης γίνονται σε τρεις χώρες που δεν είναι ε, χώρες που παράγουν πολλά αυτοκίνητα. Στο Λουξεμβούργο έγιναν χίλια τεστ μεταξύ 9 και 14 επιχειλίων οχημάτων και στην Ολλανδία αλλά και στη Μάλτα Όπως λέτε στην απάντησή σας ε, στην ερώτηση 2, λέτε ότι αυτό συνέβη γιατί οι συνθήκες που ισχύουν στα κράτη-μέλη δεν είναι όλες εξίσου αυστηρές. Ποιες ε, διαφορές υπάρχουν ε, στις τιμές, στις παραμέτρους. Εφαρμόζονται για τα διάφορα εθνικά τεστ. Και επιπλέον ποιες ενέργειες ε, αναλάβατε αυτά τα χρόνια γιατί από ό,τι βλέπω στις διάφορες εκθέσεις ότι τα, τα αυτοκίνητα βέβαια κινούνται, πηγαίνουν μια χώρα του βορρά και πάνε στον νότο για να κάνουν τα τεστ από την Ανατολή στη Δύση. Και το γενικό τεστ, ε, για παράδειγμα, τη μηχανή γίνεται σε μία χώρα και το τεστ των εκπομπών γίνεται σε άλλη χώρα. Τι ενέργειε κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα θέματα όλα αυτά τα χρόνια. η Επιτροπή. Οι εκθέσεις γίνονται σε χώρες... Συγγνώμη, η... αυτό που είπατε ότι οι εκθέσεις δεν γίνονται στις χώρες που παράγουν αυτοκίνητα δεν ε, ισχύει και τόσο πολύ. Ναι, μεν ε, στο Λουξεμβούργο έγιναν τα περισσότερα, αλλά η δεύτερη χώρα που πλευρά αριθμού τεστ είναι η Γερμανία που παράγει αυτοκίνητα. Βεβαίω τώρα. Είπα Λουξεμβούργο, όχι Γερμανία. Είπα Λουξεμβούργο. Ε, ε, γι' αυτό ανέφερα μόνο το Λουξεμβούργο, για τη Γερμανία, ναι. Αλλά είπατε, λέει ο πρόσωπο τη Κομισιόν, ότι εκθέσει γίνονται κυρίω από χώρε που δεν παράγουν αυτοκίνητα. Σε αυτό αντέδρασα. Γιατί η Γερμανία εξεπώνησε έκθεση και έκανε πολλές, ε, πολλά τεστ έγκρισης. Αλλά το Λουξεμβούργο και παρόμοια κράτη-μέλη κάνουν πολλές εκθέσεις για λόγους διάφορους που μπορώ να σας εξηγήσω. Πρώτα απ' όλα ε, ο τρόπος οργάνωσης των κέντρων ελέγχου. Ορισμένα κέντρα τεχνικού ελέγχου χρηματοδοτούνται με βάση τον αριθμό εγκρίσεων που ε, παράγουν. Το Λουξεμβούργο και η Μάλτα, τα δύο κράτη-μέλη που αναφέρατε, βέβαια θα πρέπει να απαντήσουν τα ίδια αναλυτικά, αλλά σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη-μέλη καθορίζουν πού θα γίνει ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο φορέας που θα χορηγήσει την έγκριση. Η Κομισιόν δεν μπορεί να παρέμβει. Και η νομοθεσία δεν προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τον ορισμό του φορέα που θα κάνει τον έλεγχο. Σε ορισμένε περιπτώσεις ή στι περισσότερες οι αρχές έγκρισης τύπου δεν είναι αυτές που κάνουν τα τεστ. Τα τεστ τα κάνουν διάφορα κεντρικά ε, και κέντρα τεχνικού ελέγχου που μπορούν να είναι ιδιωτικά, μπορεί να είναι μισοϊδιωτικά, μισοδημόσια και σε ορισμένε περιπτώσει μπορεί να είναι και σε άλλο κράτο μέλο από την αρχή έγκριση τύπου. Γι' αυτό ορισμένε αρχέ έγκριση τύπου δίνουν πολλέ εγκρίσει με περιορισμένου πόρου. Αλλά τροποποιούμε διαδικασία για να ενισχύσουμε το ρόλο των κέντρων τεχνικού ελέγχου και τις αρμοδιότητες των φορέων έγκρισης τύπου και η Κομισιόν θα μπορεί να κάνει τα δικά της τεστ και να συμμετάσχει σε άλλα τεστ. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε λέει Πρόεδρος και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις. Ο κύριος Γερμπράντη. Θα είμαι πολύ σύντομος λέει ο κύριος Γερμπράντη. Επανέρχομαι στον κανονισμό του 2008 για την έγκριση τύπου. Στο προηγούμενο μου ερώτημα ρώτησα για το αν είναι απαραίτητο οι κατασκευαστές να δίνουν πληροφορίες για τα συστήματα ανακυκλοφόρησης καυσαέριων. Το ίδιο όμως το άρθρο 3 αυτού του κανονισμού λέει και παραθέτω ετήσει της Κομισιόν οι αρχές έγκρισης τύπου θα δώσουν πληροφορίες για την ε, αποτελεσματικότητα των συστημάτων για τη μείωση των εκπομπών οξυδίων του αζότου σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται τυχαία. Υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος. Η Κομισιόν επί τη βάση όλων των πληροφοριών που είχε λάβει, όπως διαβάσαμε χθε στο Guardian, η Κομισιόν χρησιμοποίησε ποτέ αυτό το άρθρο σε σχέση με, την, με τον κανονισμό έγκρισης τύπου για το 2008. Του 2008 μάλλον. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκε αυτή η διάταξη. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να το ελέγξουμε και σας στείλουμε κάποια επιβεβαίωση έγγραφη αυτής της ε, απάντηση. Ναι, παρακαλώ. Το περαιτέρω ερώτημα μου ήταν το εξή. Στην απάντησή σας στο ερώτημα 8 είπατε ότι το 2012 η Κομισιόν έστειλε επιστολές σε όλα τα κράτη-μέλη τονίζοντας την ανάγκη να ενισχυθεί ο μηχανισμός ε, εποπτείας της αγοράς και να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη-μέλη θα τις απαραίτητες κτλ. κτλ. Υπήρχε ένα συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο να απεστάλλει αυτή η επιστολή, όπω φαντάζομαι. Και αν ναι πώ ανταποκρίθηκαν σε αυτό τα κράτη-μέλη και αν η Κομισιόν έδωσε κάποια συνέχεια σε αυτό το θέμα επί τη βάση των απαντήσεων των κρατών μελών μετά και το 2012. Το γράμμα αυτό έγινε για την, μετά από τις συζητήσεις που ετέθηκαν, που έγιναν μάλλον, για την ε, αποτελεσματική χρήση των ε, μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. Υπήρξαν ορισμένα κράτη τα οποία απίδησαν και έδωσαν ε, πληροφορίες για τις πρακτικές λεπτομέρειες της εποπτείας της αγοράς που ασκούν. Μία από τις συνέπειες αυτής ε, της ε, επιστολής είναι οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν. Οι εργασίες που ξεκίνησαν για να τροποποιηθεί ριζικά το βασικό κείμενο σε ό,τι αφορά την ένδυση τύπου το 2046, γιατί φάνηκε ότι το κείμενο αυτό το αρχικό δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες εποπτείας της αγοράς, δεν έδινε τις απαραίτητες ε, ε, λεπτομέρειες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια. Κύριο Στουριδάκη. θα κάνω εγώ μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στο θέμα αυτό. Όλοι μιλάνε για την Κομισιόν. Εγώ θα ήθελα, επειδή θα μας ζητήσουν να μας πούνε και οι εκλογές μας, ποιος ήταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο πρόεδρος Σούλτς, ο οποίος ε, ήταν και αυτούς που πίεσαν για την ε, δημιουργία αυτής της ε, Επιτροπής. Εγώ δεν θυμάμαι τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια σε καμία περίπτωση να υπάρχει μια υπόμνηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Ίσως μπορείτε να με πληροφορήσετε καλύτερα εσείς. Δεν θα σας ρωτήσω βέβαια εσάς για τις πολιτικές δραστηριότητες του κυρίου Σούλτς, αλλά θα ήθελα να ξέρω αν εσείς είχατε προειδοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την, την ε, διαδικασία της εκπόνησης έκθεσης CARS 2020, αν υπήρξε μια προφορική ερώτηση ή κάτι άλλο από το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά και αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσεκλήθη να συμμετάσχει στη συνάντηση των CARS 2020, συνάντηση υψηλού επίπεδου, που με πρόταση του Επιτρόπου Ταγιάννη ε, απέριψε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απέριψε την παρουσία του του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχετε κάποια λεπτομέρεια για αυτή τη συνάντηση. σε πολλά επίπεδα. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ρωτήσετε γιατί δεν θέλησε να συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση ΚΑΣ 2020. Μετά από τις εργασίες της ΚΑΡΣ 2020 υπήρξε μια ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο και η οποία ήταν και αντικείμενο συζητήσεων και ενός ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη στρατηγική για τις εκπομπές και την ε, μέτρηση σε πραγματικές συνθήκες και την στρατηγική για την εποπτεία της αγοράς Όλα αυτά περιλαμβανόντουσαν στην ανακοίνωση της Κομισιόν και συζητήθηκαν όταν ενεκρίθηκε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι μπορώ να κλείσω εδώ. με τα στοιχεία αυτά που μας δώσατε έχουμε νέα στοιχεία για την ε, έλλειψη δράση από τα κράτη-μέλη και της Κομισιόν. Γι' αυτό θέλω να θέσω τρία ερωτήματα. Πρώτον, κατά τη διάρκεια αυτής της ε, ε συνάντησης φάνηκε ότι υπήρχαν τρία μπλοκ χωρών που ζητούσαν ταχύτητα, όπως η Δανία, για την εφαρμογή του RDE. Υπήρχαν άλλες που θέλανε περισσότερο χρόνο και κάποιες είχαν ε, προβάλλει προσκόμματα. Ποιε ήταν οι χώρε που προέβαλαν προσκόμματα κατά τη διάρκεια αυτή τη συνάντησης. Α, τέτοιου είδου πληροφορίε μπορεί να σας δοθεί από την Κομισιόν μόνο ε, υπό, την, τον όρο της εμπιστευτικότητας, λέει ο κ. Κασίγου. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, τι εμπιστευτικότητα μπορεί να υπάρχει όταν ε, αναφέρατε ότι κάποιοι ήταν ε, πρόθυμοι και αναφέρατε, κάποιοι άλλοι ήθελαν χρόνο και αναφέρατε, άρα και για την τρίτη κατηγορία πρέπει να μας αναφέρετε. Τώρα άλλη ερώτηση. Στη συνεδριάση της Τεχνικής Επιτροπής κανένα κράτος μέλος δεν προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτοί οι μηχανισμοί αλλίωσης που θα μπορούσε να υποπτεύεται ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από κάποιους από τους κατασκευαστές. δεν έχω καμία γνώση τέτοια. Από ό,τι ξέρω, κανείς ποτέ, λέει η Κομισιόν. Τρίτον, θα μπορούσατε παρακαλώ να μας ε, κοινοποιήσετε τα πρακτικά αυτών των συνεδριάσεων της Τεχνικής Επιτροπής. Αυτό είπα και προηγουμένως. Εμείς δίνουμε αυτά τα πρακτικά μέσα στα πλαίσια της Συμφωνίας Εμπιστευτικότητος που έχει συζητήθει μεταξύ της Κομισιόν και ημών με ύψιλον. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα έγγραφα αυτά θα είναι διαθέσιμα είτε στην αίθουσα εμπιστευτική ανάγνωσης ή αλλού. Θα γίνουν διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά. Αύριο, αύριο, σήμερα τα μου θα συνεδριάσουν οι συντονιστέ και θα σα πούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Έκανα αυτές τις δύο ερωτήσεις και έχω τώρα μια τρίτη συνδεόμενη ερώτηση. Πρώτον, ποιες χώρες ε, έθεσαν προβλήματα. Δεν μου είπατε. Δεύτερον, αν υπήρξε κάποια ανακοίνωση στην Τεχνική Επιτροπή, δεν μου είπατε κάτι τέτοιο. Εμένα η τρίτη μου ερώτηση είναι, δεν σας είναι εκπληκτικό ότι μετά από το σκάνδαλο σε δέκα μέρες μπόρεσαν να, να εφαρμοστούν όλα αυτά. Μήπως ε, εσείς είχατε κάποιες υποψίες επομένως. Ναι. Κύριε Ντάλη. Σας ευχαριστώ. Σας παρακολούθησα με προσοχή από την αρχή και υπάρχει κάτι το οποίο με εκπλήσει. Λέτε ότι υπήρχαν υποψίες για τη χρήση λογισμικού που οδηγούσε σε χειραγώγηση πριν από το σκάνδαλο της ε, Volkswagen. Βέβαια δεν είχατε κανένα συγκεκριμένο ε, παράδειγμα, κανένα όχημα το οποίο να σας δημιούργησε υποψίες. Αυτά όμως που λένε τα πρακτικά του εργαστηρίου σας το 2010 για την νομοθεσία στα θέματα αυτά λέγεται εκεί πέρα ότι ένα αυτοκίνητο το οποίο δοκιμάστηκε έδειξε μια τεράστια α, απόκληση σε σχέση με τα όρια που προβλέπονται όταν έγινε ο έλεγχος σε χαμηλή θερμοκρασία. Μήπως όμως θα μπορούσατε ήδη από τότε να θεωρείτε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Και τι έγινε αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν που είχατε δοκιμάσει, τι το κάνατε πήρατε τηλέφωνο τον κατασκευαστή, ζητήσατε να μάθετε από τις εθνικές αρχές για να καταλάβετε γιατί αυτό το αυτοκίνητο μπόρεσε να έχει τόσο μεγάλες αποκλήσεις. Τι κάνατε για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Ε, νομίζω ότι ήταν το πρώτο θέμα για το οποίο απάντησα το με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε σήμερα και στο άρθρο ε, που δημοσιοποιήθηκε χθε ήταν ένα βερζινοκίνητο. που είχε μια πολύ μεγάλη εκπομπή οξυδίων του αζότου σε ε, συγκεκριμένο στάδιο της δοκιμής Euro 6 το οποίο είναι φυσικό φαινόμενο και δεν μας εξέπληξε. Και επίσης ήταν κάτι το οποίο προβλέπεται από τις εξαιρέσεις του κανονισμού. Επομένως δεν μας δημιούργησε την υποψία αυτό το αποτέλεσμα της μέτρησης ούτε θα μπορούσε να χρησιμοποιείται μια διάταξη αναστολής. Για αυτό που υπονοείται ότι χρειάστηκε ένα σκάνδαλο για να ε, υιοθετηθεί νομοθεσία πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν ισχύει. Είχαμε ξεκινήσει την α, επεξεργασία του πακέτου RDE τον, Οκτεύ, τον Οκτώβριο και αυτό υιοθετήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Η συζήτηση μάλλον ξεκίνησε τον Οκτώβριο και εγκρίθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η προετοιμασία είχε ξεκινήσει πολύ πριν. Ευχαριστώ. Κύριε Βουλευτής. Ναι, αλλά είπατε κάτι το οποίο εγώ βρίσκω σκανδαλώδες, ότι αυτό το λογισμικό, οι ε, διατάξει αναστολή, εκείνη την εποχή δεν ήταν η προτεραιότητά μα. Έτσι είπατε πριν. Επίση, χρειάστηκαν 10 χρόνια για να εφαρμοστεί η νομοθεσία του 2007, με άμεσες επιπτώσεις για την προστασία του καταναλωτή και την υγεία του πληθυσμού. Και θέλω να καταλάβω κάποια στιγμή τι είναι αυτό που προκαλεί αυτή την καθυστέρηση. Τι φταίει και νομοθεσία που υιοθετείται το 7, φτάνουμε το 2017 και δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Και αυτό είναι δικιά σας ευθύνη ως ε, θεματοφύλακες των συνθήκων να μας εξηγήσετε γιατί δεν εφαρμόζεται νομοθεσία. Η απάντηση της Επιτροπής. Η χρήση τέτοιου λογισμικού απαγορευόταν. Επομένως είχε αναλυφθεί δράση σε αυτόν τον τομέα. Μετά, όπως είπαμε, είχε αναγνωριστεί ότι υφίσταται ο κίνδυνος, γιατί ξέραμε ότι υπήρχε αυτό το λογισμικό, αλλά δεν είχαμε αποδείξεις ότι σε κάποιο συγκεκριμένο όχημα είχε χρησιμοποιηθεί. Και γι' αυτόν τον λόγο ασχοληθήκαμε με αυτό που κατά την άποψή μας ήταν το πιο σημαντικό, δηλαδή να αναπτυχθούν τεστ, ε, συστήματα μετρήσεων, ε, πιο αποτελεσματικά και ασχοληθήκαμε αν θέλετε με το δομικής φύσεως ζήτημα και όχι με το λογισμικό. Ευχαριστώ. Και εγώ πρέπει να πω ότι ε, δεν είμαι με τους πολύ απογοητευμένους, αλλά θέλω να καταλάβω καλύτερα πώς εργάζεστε. Είχατε μια ερώτηση προηγουμένως για το που υπάρχει σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας για τους μηχανισμούς. Και είπατε ότι δεν γνωρίζατε. Και είπατε ότι προχωράει αυτή η προσπάθεια τώρα. Έχουμε όμως κάποια κείμενα από κάποιους φορείς, όπως για παράδειγμα το Διεθνές Συμβούλιο για Καθαρή Κυκλοφορία και ξέρετε ότι οι Αμερικανοί προηγούνται. Πώς λειτουργεί στο εσωτερικό της Κομισιόν, τα διαβάζετε αυτά που γράφουν άλλοι ή δεν σας απασχολούν τι συμβαίνει αλλού. Δεν θεωρείτε ότι είναι δουλειά σας να κάνετε συγκρίσεις με αυτά που γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου. Όπως είπα και νωρίτερα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των νομοθεσιών ε, στις ΗΠΑ και τη δική μας. Απλώς, στη μία περίπτωση, στις ΗΠΑ ήταν υποχρεωμένοι να δηλώνουν τη στρατηγική ελέγχου των εκπομπών τους, ενώ εμείς ε, δεν είχαμε αυτή την υποχρέωση. Και η επιτήρηση της αγοράς στις ΗΠΑ είναι πιο ομοιόμορφη από ότι στην Ένωση. Γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν θέλει να συμπληρώσει κανείς. Κάτι ακόμη. Ε, το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ αυστηρό, πολύ πλήρες. Άρα, παρά, αλλά παρά το ότι είχαν ε, αυτό το σύστημα ε, ε, τόσα χρόνια, δεν αποκάλυψε το μηχανισμό αυτό ο περιβαλλοντικός φορέας τους. Χρειάστηκε πολύς χρόνος και ούτως ή άλλως το συζητάμε ε, από το 2014. Άρα ε, αξιοποιούμε τις καλές πρακτικές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες του, όσο καλό και αν φαίνεται. Η κυρία Κόστιγκερ. Μία δεύτερη ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες ε, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από το σώμα μας. Πώς αντιμετωπίζετε ως υπηρεσίες της Κομισιόν τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Είναι μόνο επιφανειακές οι απαντήσεις σας ή το ψάχνετε σε βάθος. Έχετε μήπως ε, μία στάνταρ απάντηση ακόμη και αν αναφέρονται συγκεκριμένες υπόνοιες ή δεν γνωρίζετε πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι ερωτήσεις. Η Κομισιόν. Προφανώς οι προφορικές ερωτήσεις αντιμετωπίζονται με μεγάλη προσοχή και αν υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές, συγκεκριμένα στοιχεία, τότε τα ελέγχουμε. Αν οι ερωτήσει εκφράζουν γενικέ και αόριστες ανησυχίε, ε, τότε προφανώς ε, το εξετάζουμε, αλλά έχει να κάνει με το πώς διατυπώνεται η κάθε ερώτηση και τι περιέχει. Από αυτό εξαρτάται πώς αντιμετωπίζεται. Ο κύριος Χένκελ. Μερικές σύντομες ερωτήσεις. Από πότε ξέρετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1998 ήδη υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, μια τέτοια υπόθεση για κάποιον κατασκευαστή φορτηγών. Κομισιόν. Μόλις ε, μάθαμε γι' αυτό, ξεκινήσαμε κι εμείς το 98, ε, ε συμπεριλάβαμε την απαγόρευση αυτού του μηχανισμού σε ένα νομοθέτημα το 98. Ο κ. Χένκελ συνεχίζει. Είπατε προηγουμένως ότι ο ορισμός του λογισμικού που χρησιμοποιείται είναι εντάξει. Αλλά η εφαρμογή της διάταξης που περιέχει αυτόν τον ορισμό ήταν ελαττωματική, αν σας κατάλαβα καλά. Αυτή τη στιγμή κατηγορούνται όμως και η Fiat και η Opel ότι χρησιμοποιούν μία ε, αρκετά διευρυμένη και γενναιόδορη ερμηνεία αυτού του ορισμού. Μήπως θα έπρεπε να διευκρινιστεί ο ορισμός, για παράδειγμα, για το φάσμα θερμοκρασιών κομισιών. Επαναλαμβάνω, η νομοθεσία είναι σαφής. Ίσως να υπάρχει ανάγκη εναρμονισμένης εφαρμογής της νομοθεσίας. Και η Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια. Μπορούμε να δώσουμε συμβουλές και κατευθύνσεις. Αλλά για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε αναλυτική πληροφόρηση. Το είπα και προηγουμένως. Δεν την έχουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε αναλυτικά, αναλυτικά στοιχεία για τα αποτελέσματα των τεστ, τι απεκάλυψαν, για να μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε την νομοθεσία με βάση τα στοιχεία. Αυτά είμαστε διατεθειμένοι να τα κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε εν κενό. Αυτή τη δυσκολία έχουμε. Εν τω μεταξύ, λέει ο κύριος Χένκελ, θα ακούσατε τι γίνεται στην Ιαπωνία. Η Σουζούκη και η Μιτσουμπίση. Φαίνεται ότι έχουν διαφορετικούς τρόπους για να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των τεστ. Δεν χρειάζεται να βάλετε νέο ε, λογισμικό. Μπορεί να, ε, για παράδειγμα, να στέλνετε αυτοκίνητα πιο ελαφρά για τα τεστ. Πώς θα κλείσετε όλες αυτές τις τρύπες στην νομοθεσία. Κομισιόν. Νομίζω ότι οι δοκιμασίες αντί σε πραγματικές συνθήκες, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μπορούν να εμποδίζουν τη χρήση διατάξεων αναστολής. Γνωρίζετε ότι είμαστε η μόνη περιοχή του κόσμου που θα χρησιμοποιήσουμε δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις ε, ατασταλίες ή τι απάτε, Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε για το Ε, δεν εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο με φορητές συσκευές μέτρησης και βρισκόμαστε τώρα στη φάση αυτή παρακολούθησης. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα PEN στον πρώτο χρόνο και μετά θα εξετάσουμε την εφαρμογή των κανόνων. Αν υπάρξει κάτι το οποίο έρθει στην προσοχή μας, το οποίο θα μας κάνει να ξανασκεφτούμε για τη βελτίωση, θα το κάνουμε. Είναι μια διαδικασία λοιπόν εν εξελίξει. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν και δεν θα πούμε ότι εφόσον εφαρμόζεται αυτό το σύστημα τελείωσε η διαδικασία. Στην απάντησή σας στο ερώτημα 10 λέτε ότι η Κομισιόν έχει κατ' επανάληψη ζητήσει από τα κράτη-μέλη να δώσουν τα στοιχεία των εθνικών ε, ερευνών σε σχέση με τις ε, με τις εκπομπές των ε, οχημάτων. Είπατε ότι μέχρι στιγμής έχει μόνο από την ε, Γερμανία, την Αγγλία και την Γαλλία. Τι έχει όμως κάνει η Κομισιόν μετά από αυτή την άρνηση των άλλων κρατών να δώσουν στοιχεία. Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο αυτά τα περιορισμένα στοιχεία η Κομισιόν στη συνέχεια. Αν υπάρχει δισταγμός των κρατών μελών, σίγουρα δεν υπάρχει άρνηση να διαβιβάσουν στοιχεία. Ζητήσαμε την διαβίβαση των στοιχείων αυτών από την Κομισιόν. Η Επίτροπος μας έκανε μια αίτηση, 7 Ιουνίου την επανέλαβε αυτή την αίτηση. Θα δούμε τι θα γίνει. Εάν δεν υπάρξουν απαντήσεις, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε τις δυνατές μας αντιδράσεις. Τούτου λεχθέντος όμως, επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή της ακρόασης ότι όσο δεν έχουμε αυτές τις πληροφορίες, εμείς δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε τα συμπεράσματα των εκθέσεων των τριών αυτών χωρών που έδωσα στοιχεία. Αυτό σημαίνει όταν λέτε ότι θα χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες, τι θα κάνετε συγκεκριμένα, τι εννοείτε ακριβώς, αν δεν πάρετε τα στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Δεν θέλω να επεκταθώ για το θέμα αυτό, αλλά η Κομισιόν θα πρέπει να εξετάσει τα περαιτέρω βήματα. Ένα δεύτερο ερώτημα τώρα έχω να σας θέσω. Στην γραπτή σας απάντηση στην ε, ερώτηση 5 για τα onboard diagnostic, diagnostic systems. Είπατε ότι τα στοιχεία των OBD στην Ευρώπη δεν συγκεντρώνονται συστηματικά. Ενώ αντίθετα στι ΗΠΑ υπάρχει υποχρέωση τα στοιχεία αυτά να δίδονται στι αρμόδιε αρχέ. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση και αν θεωρείτε ότι είναι σωστή αυτή η διαδικασία, δεν θεωρεί ότι υπάρχει αξία, προσθέμενη αξία από την Κομισιόν στη χρήση αυτών των στοιχείων OBD και ποια συμπεράσματα θέλετε εσείς να αντλήσετε από αυτή τη διαφορά που υπάρχει. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι δεν μπορώ να σας πω ποια είναι, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουμε διαφορετικούς κανόνες από τους δεσμευτικούς κανόνες στις ΗΠΑ. Αυτές τις πληροφορίες φυσικά συλλέγονται από τις ε, κατασκευαστικές εταιρείες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πληροφορία. Το ερώτημα τώρα είναι τι είδους πληροφορίες θα ήταν χρήσιμες για την Κομισιόν, γιατί φυσικά δεν είναι όλες οι πληροφορίες οι οποίες θα επιτύχουν το στόχο που έχουμε, είναι να, δηλαδή να δούμε τα προβλήματα με τις ε, εκπομπές. Κοιτάμε τώρα μήπως υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε αυτούς τους κανόνες και αυτό είναι μια συνεχής διαδικασία. Ο κύριος Σούτσε. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί, αλλά φοβάμαι ότι πρέπει να τα επαναλάβω γιατί δεν ήταν σαφή η απάντηση. Εγώ είμαι μηχανικός, δεν είμαι νομομαθής και έχω ένα πρόβλημα με το αν διατυπώνω τα πράγματα με τέτοια ασάφεια. Θέλω να επανέλθω λοιπόν σε ένα ζήτημα, τον ε, κύκλο NEDC, ε, τον Ευρωπαϊκό Κύκλο Δοκιμασιών. Έχετε πει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική, πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης, αλλά στον κανονισμό του 2007 στο άρθρο 5.1 λέει ότι ένα σύστημα μείωση των εκπομπών πρέπει να ανταποκρίνεται σε πραγματικέ συνθήκε. Μα δεν ορίζει κανεί ποιες είναι αυτέ οι πραγματικέ συνθήκε. Τι σημαίνει για σα φυσιολογικές συνθήκε οδήγηση. Εσεί εξακολουθείτε όμω να κάνετε όλα αυτά τα οποία γίνονται μόνο στο εργαστήριο και δεν λαμβάνετε υπόψη πραγματικέ συνθήκε. Ποια είναι η απάντησή σα σε αυτό. Σίγουρα δεν είναι σαφής η, το τι είναι φυσιολογικές συνθήκες οδήγησης. Αυτό φυσικά σημαίνει το σύνολο των δυνατοτήτων οδήγηση στον πραγματικό κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να καταμετρηθούν όλα αυτά και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε τους παράγοντες συμμόρφωσης, τους συντελεστές συμμόρφωσης μέχρι να αναπτύξουμε δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες. Όπως ε, είπα όμως προηγουμένως, η νομοθεσία υποχρεώνει την Κομισιόν να ε, θεσπίσει μια μέθοδο, ε, μια μέθοδο μέτρησης. Μέχρι τώρα αυτό σήμαινε μέτρηση σε εργαστήρια. Τώρα το τροποποιούμε αυτό, θα προχωρήσουμε στις δοκιμασίες σε πραγματικές συνθήκες, αλλά όταν εκδόθηκε αυτός ο κανονισμός, εμείς προχωρήσαμε σε δεσμευτικές ε, μετρήσεις στο εργαστήριο, που δεν έρχεται σε αντίφαση με το πνεύμα του κανονισμού. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνετε τώρα ή τι θα κάνετε σε μερικού μήνε ή σε μερικά χρόνια και τι θα γίνει στη συνέχεια. Υπάρχει ήδη ένα τεράστιο ερωτηματικό που θα πρέπει να θέσουμε για τη χρήση των εργαστηριακών ε, δοκιμασιών. Τώρα, πώ κρίνετε εσεί επίση την τεχνική ικανότητα των ε, φορέων της Κομισιόν Φυσικά οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι άλλοι εμπλεκόμενοι στον τομέα αυτό έχουν πραγματικά πολύ ψηλέ γνώσει στον τομέα αυτό των ε, αυτοκινήτων. Η Κομισιόν έχει τι απαραίτητε εμπειρογνωμοσύνε για να σταθεί στο ύψο των προκλήσεων. Εμεί έχουμε κάθε εμπιστοσύνη στην τεχνική ικανότητα των συναδέλφων μα είτε στην DG Grow, στην DG Κλίμα και, στα, στο και κοινό κέντρο ερευνών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, τούτου όμω λεχθέντο εμείς βασιζόμαστε και σε εμπειρογνωμοσύνη από τα έξω, όπως ανέφερα προηγουμένως από τα κράτη-μέλη, από, τους, από τα πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ. Δεν έχουμε λοιπόν έλλειψη ε, εμπειρογνωμοσύνης που μπορεί να συμπληρωθεί από εξωτερικές πηγές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στη διάθεσή μας. Currents. Και εγώ σας ευχαριστώ κατάλαβα από τις προηγούμενες απαντήσεις ότι εσείς δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι υπήρξε ε, προσπάθεια εμποδισμού από κράτη-μέλη, από άλλους φορείς, γιατί χρειάστηκε πάρα πολύ καιρό για να μπορέσουν να θεσπιστούν αυτές οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Υπάρχει όμως το θέμα της λογοδοσίας. Στις Ηνωμένες, στην Σοβιετική Ένωση ξέραμε ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ήταν αναποτελεσματικό. ή μηχανική φτιάχνανε τους, τους, ε, τις προδιαγραφές για να φτιάξουν μια γέφυρα, αλλά μετά όλοι κλέβανε στα υλικά. Οπότε κανείς δεν ήξερε αν θα λειτουργήσει η γέφυρα ή όχι. Αλλά είχαν έναν τρόπο να το κάνουν αυτό, να δοκιμάσουν. Παίρνανε ένα φορτηγό, το γεμίζαν χαλί, παίρνανε φορτηγά γεμί, γεμάτα χαλί και τα βάζαν στη γέφυρα και αν η γέφυρα δεν έπεφτε τότε ήταν ασφαλής. Βέβαια, λένε, έχω δει σε έντυπα ότι στις ε, χώρες της ε, στις βόρειες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν ε, σε, σε εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτομάζες ότι οι διευθυντές του εργοστασίου πίνουν το νερό για να δουν αν ασφαλές. Ποιος όμως θα αναπνεύσει τα καυσαέρια για να ξέρουμε την είναι ασφαλή. Ποιος θα αναλάβει να είναι υπόλογος για τα θέματα αυτά και πότε θα το ε, ε, εξασφαλίσετε αυτό. Οι δοκιμασίες οι οποίες έχουν εισαχθεί θεωρούνται από την Κομισιόν και τα 28 κράτη-μέλη ότι είναι ε, επαρκή για να ανακλούν τις πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης χρήσης των οχημάτων και φυσικά θα μπορούν και οι εμπλεκόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν τεστ για να δουν αν οι στόχοι οι οποίοι έχουν διατυπωθεί πράγματι εκπληρώνονται στην πραγματικότητα. Θα υπάρξει ένα τέτοιο είδους ελέγχο. Κανείς βέβαια δεν θέλει να είναι ο οδηγός του φορτηγού που είναι γεμάτο με χαλίκι. Ναι, αλλά για να δώσω συνέχεια σε όλα αυτά. Λέτε όλοι ότι αυτές οι δοκιμασίες είναι επαρκείς. Με ποιο τρόπο όμως μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πράγματι επαρκείς οι δοκιμασίες, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απόλυτα θεωρητικό επίπεδο. Δεν είμαστε το 2017. Τι θα πρέπει να αλλάξει στο σύστημα για να το κάνει πιο αξιόπιστο, πώς θα ξέρουμε ότι θα είναι αξιόπιστες αυτές οι οι αλλαγέ. Από τις αρχές του χρόνου για λόγους εποπτείας έχουμε εισαγάγει αυτές τις ε, δοκιμασίες πρωτού γίνουν υποχρεωτικές το 2017. Δηλαδή ήδη τώρα παρακολουθούμε τι τις δοκιμασίες αυτές και τα αποτελέσματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να λειτουργούν αυτέ οι δοκιμασίε και θα υπάρξει συνέχεια στη, μετά το 2017 γιατί όπω ξέρετε από το 2017 η πρόθεση είναι να υπάρχει ετήσια επισκόπηση των παραγόντων συμμόρφωσης για να δούμε αν μπορούν να μειωθούν γιατί η εμπειρία μας με τα τεστ θα αυξηθεί και ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των παραγόντων συμμόρφωσης. Η διαδικασία λοιπόν παρακολούθησης και βελτίωσης έχει ήδη ξεκινήσει. Τέλος, τελευταία ερώτηση. Η κυρία Μπονιφά. Όχι, όχι, κλείνουμε λέει η πρόεδρος. Συγγνώμη, Κλοντ, όλοι έχουν ξεπεράσει το χρόνο τους και είμαστε στο τέλος του χρόνου της συνεδρίασης. Κύριος Τέρμες χωρίς χρόνο. Όχι, Κλοντ. Λυπάμαι, Κλοντ. Αν είχαμε χρόνο, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Τούρμες. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Κύριε Μπονιφά. Στο πρώτο παράπτυμα που μας έστειλε η Επιτροπή, στη δεύτερη σας απάντηση, αναφέρεται ποιες ήταν οι προτάσεις της CEA στις οποίες δεν συμφωνήσατε η ε, Ένωση τη αυτοκινητοβιομηχανιών λοιπόν, τη μείωση τη ταχύτητα, αυτό δεν έγινε δεκτό. Και το δεύτερο ήταν η εκκίνηση του κινητήρα από την ψυχρού κινητήρα και επίση το να μετρούνται οι εκπομπέ τρία λεπτά μετά από την εκκίνηση του κινητήρα. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, ποια ήταν τα στοιχεία τα οποία ζήτησε η αυτοκινητοβιομηχανία να ε, συμπεριληφθούν, μια και όπω σωστά μα είπατε συμμετέχουν οι εμπειρογνώμονε αυτοί ε, στις συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να σας στείλουμε συμπληρωματικές πληροφορίες, επιπρόσθετες, σε σχέση με αυτά που σας στείλαμε στο παράτημα 1, το οποίο θα σας δείχνει ακριβώς πώς κατέληξε στην θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς μετά συζητήθηκαν αυτά τα θέματα στην τι συμβεί. Ο στόχος πάντα ήταν να επιτευχθεί η απαιτούμενη ειδική πλειοψηφία στη TCMV. Δεν είχαμε επιδίωξη να ικανοποιήσουμε καμία ομάδα πίεσης της αυτοκινητοβιομηχανίας ή άλλη Μπορούμε λοιπόν να σας αποστείλουμε περισσότερα στοιχεία για το σκεπτικό, για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να υπάρξει συμφωνία στη τι συμβεί. Μπορώ να έχω τουλάχιστον μία απάντηση γιατί αλλάξατε αυτό το όριο ταχύτητας τουλάχιστον αυτό και επίσης γιατί δεν δεχτήκατε να υπάρχει και, ο, και η δοκιμή, η μέτρηση σε υψηλή ταχύτητα, η απάντηση της Επιτροπής. Εγώ θα σας απαντήσω για την εκκίνηση ε, από, με ψυχρό κινητήρα. Εμείς σκοπεύουμε στο νέο πακέτο αντί e να το συμπεριλάβουμε αυτό, στην, στο νέο πακέτο νομοθεσίας, και ο λόγος που αυτό δεν μπορούσε να γίνει πιο νωρίς ήταν γιατί χρειαζόταν χρόνος ε, για να έχουμε τις τιμές αναφοράς που θα μας επέτρεπε να συγκρίνουμε αυτά τα στοιχεία. Δεν το κάναμε για να ικανοποιήσουμε την αυτοκίνητο βιομηχανία. Αυτό είναι από τα παραδείγματα, ένα παράδειγμα από αυτό που αναφέρατε και θα σας απαντήσουμε στα υπόλοιπα γραπτός. Η Πρόεδρος, ξέρετε ότι προσπαθώ να χειριστώ το χρόνο έτσι ώστε να έχουν όλη τη διάθεση, χρόνο στη διάθεσή τους να υποβάλουν ερωτήσεις. Δίνω ένα λεπτό. Τώρα που έχουν προταθεί τα πέμψη, πώς θα εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει κολλησιεργία στην ομάδα εμπειρογνωμόνων και πώς δεν θα χάσουμε άλλα δύο χρόνια. Όταν εσείς οι ίδιοι μας λέτε ότι οι αντιπροτάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στην πραγματικότητα προσπαθούν να ροκανίσουν το χρόνο. Το τι έγινε το 2012-2013 2011 ε, μέχρι και 2013 μπορείτε να το βρείτε στην έκθεση του 2013. Όλα τα συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Δεν μπορώ να αξιολογήσω εδώ αν ήταν γρήγορο ή αργό, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σας αναφέραμε όλα όσα έγιναν. Σεπτέμβριος του 2013, δημιουργία μιας task force, μιας ομάδας εργασίας και θα σας ρωτώ αφού θα έπρεπε να ολοκληρώσει εργασίες τη μέχρι το μέσο του 2014 που βρισκόμαστε. Δημιουργήθηκε η πρόεδρος. Ε, είχαμε πει ένα λεπτό σας έδωσε το λόγο. Πάρε. Κλόντ, θα επανέλθουμε, λέει η πρόεδρος. Ο κύριος Βουλευτής δεν λαμβάνει όμως απαντήσεις από αυτούς τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Η ε, Πρόεδρος, θα το συζητήσουμε το ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου. Λοιπόν, Παρά την απογοήτευση που νομίζω ότι μπορέσατε να διασταθείτε από τα διάφορα μέλη τη Επιτροπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τη Επιτροπή για την πολύ ενδιαφέρουσα και ενδελεχή συζήτηση όλων αυτών των ζητημάτων. Να ευχαριστήσω του εκπροσώπου τη Επιτροπή. Είναι προφανέ ότι θα συνεχίσουμε τι συζητήσει για αυτά τα θέματα, θα ήθελα να μεταδώσετε το εξή μήνυμα στους προϊσταμένους σας και στους πολιτικούς προϊσταμένους σας ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να τους μεταδώσετε το μήνυμα ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο συνεργασίας της Επιτροπής με την Επιτροπή μας. Ε, και με το γεγονό ότι δεν έχουμε λάβει τα στοιχεία που έχουμε ζητήσει, θα πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για τι επόμενε συναντήσει. Σα ευχαριστώ.